colleghi, grazie per la presenza. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Βέβαια, ο καιρός δεν βοηθάει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την ανοιχτή ακρόαση και χαίρομαι να σας καλωσορίσω όλους. Το θέμα είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον μεταναστευτικές ροές που προκαλούνται από αιστείες αστάθειες ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η, οργανώνεται η ακρόαση σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης, προετοιμάζοντας πρωτοβουλίες περαιτέρω. Η μετανάστευση είναι ένα σφαιρικό φαινόμενο, λέω κάτι το προφανές. Ένα φαινόμενο το οποίο ακριβώς επειδή φύγει εκατομμύρια ανθρώπων πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και οικονομικά και σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται μια δημόσια ακρόαση σε συνεργασία με τη δική μας Επιτροπή. Η σημερινή συνάντηση και η πρωτοβουλία που θα ακολουθήσει με τη συνεισφορά όλων των εμπειρογνωμόνων οι οποίοι είναι παρόντες και τους οποίους θα παρουσιάσω έχει σαν στόχο να εμβαθύνει την διάσταση της εξωτερικής πολιτικής εκεί που συνδέεται με το μεταναστευτικό φαινόμενο και να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τις χώρες προέλευσης και μέσω της εξωτερικής πολιτικής της και όχι μόνο βέβαια. Είναι σαφές ότι η εξωτερική πολιτική δράση έχει σαν στόχο την δημιουργία πολιτικής σταθερότητας της χώρες προέλευσης και ενίσχυση των πρακτικών χρηστής διακυβέρνησης, κράτους δικαίου και λειτουργίας εύρυθμης των δημοκρατικών θεσμών. Αυτό θα επιτρέψει να βοηθήσουμε αποτελεσματικά μακροπρόθεσμα και να καταστήσουμε τη μετανάστευση μια δυνατότητα και όχι μια αναγκαιότητα. Αυτή η μακροπρόθεσμη στρατηγική, διαρθρωτική στρατηγική, αφορά κυρίως ε, τα μεταναστευτικά ρεύματα τα οποία δημιουργούνται λόγω πολιτικής αστάθειας. Κλείνοντας αυτή τη μικρή εισαγωγή θα ήθελα να πω ότι η ανάλυση και του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις μεταναστευτικές ροές είναι σημαντική λόγω της αναδιαπραγμάτευσης και των οικονομικών μέσων για την εξωτερική πολιτική το 2014 στα πλαίσια της αναθεώρησης της πολιτικής μας για τις χώρες γειτονίας. Έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα τον Ρομπέρτους Ρόζεμπουργκ, υπεύθυνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ανάπτυξης, τον Μπερνάρ Μπρουνέ, τμήματάρχη της εξωτερικής υπηρεσίας Ρελέξ, η Πάολα Πάτσε της Διεθνούς Οργάνωσης Μεταναστεύσεων, ο Ενρίκε Μποναβέντε, υπεύθυνο ε, του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας, και ο κύριος Φιλίπ Τεμπρουκέρ, καθηγητής στην, στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, θα έρθει όπου να είναι. Πριν δώσω το λόγο στους ομιλητές, θα ήθελα να ζητήσω από τον Αντιπρόεδρο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, που συμπροεδρεύει θα έλεγα, να θέσει το θέμα και σε σχέση με την πολιτική της ανάπτυξης. Καλημέρα σας, χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτήν την ε, από οργανωμένη συνάντηση που ψάχνει να βρει τη σύνδεση ανάμεσα στην εξωτερική πολιτική και τη μετανάστευση. Η μετανάστευση έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, αλλά τα κράτη-μέλη δεν έχουν απαντήσει στα φαινόμενα αυτά με τον κατάλληλο τρόπο, φαινόμενα τα οποία δεν φαίνεται να μειώνονται τα επόμενα χρόνια και εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους. Νομίζω ότι οι συγκεκριμένες δράσεις, σωστά στοχευμένες, μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αιτίες που προκαλούν τα μεταναστευτικά ε, κύματα, ιδιαίτερα μέσω της βοήθειας που έχει στόχο την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ευημερία. Η εξωτερική πολιτική μπορεί να βοηθήσει φυσικά και σε επίπεδο αναπτυξιακής βοήθειας. Η αναπτυξιακή βοήθεια από την άλλη από μόνη της ε, δεν επαρκεί Βασική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής είναι ακριβώς όμως η σύνδεση ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε την κινητικότητα, την δυνατότητα μετακίνησης των πληθυσμών σαν ανθρώπινο δικαιώματα, αλλά σε επίπεδο επιλογής και όχι σε επίπεδο αναγκαιότητας ή υποχρέωσης. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη και όταν έχουμε μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έχουμε μικρότερη μετανάστευση. Θα πάρω το λόγο και κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόζεμπουργκ, έχετε το λόγο 10 λεπτά περίπου. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Προβέρα και την κυρία Κρετού που έφεσαν το θέμα της μετανάστευσης σε ένα ευρύτερο ενιολογικό πλαίσιο. Πράγματι έχει φτάσει η ώρα να ξεπεράσουμε τα όρια της μεταναστευτικής πολιτικής και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με όλες τις άλλες πολιτικές μας όπως την πολιτική της ανάπτυξης. Θα ασχοληθώ με τρία θέματα. Πρώτον, Ποιοι είναι οι παράγοντες οι καθοριστικοί που πρέπει να εξετάσουμε. Δεύτερον, να δούμε τι πολιτικές κοινοτικέ είναι σχετικές με το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε και τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Όπως λέγει ο τίτλος αυτής της ακρόασης, η αστάθεια είναι θα έλεγα η βασική αιτία της μετανάστευσης. Πρέπει να κατανοήσουμε όμως τι είναι η αστάθεια αυτή. Πρέπει να το δούμε με ένα ευρύ τρόπο και όχι με περιορισμένο στενό τρόπο. Δεν μιλάμε μόνο για πολιτική αστάθεια, μιλάμε και για οικονομική αστάθεια που παίζει και αυτή σημαντικό ρόλο. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι μεγαλύτερη αιτία για τη μετανάστευση οικονομική αστάθεια. Βλέπουμε ας πούμε πρόσφυγες Βλέπουμε τον κόσμο που προσπαθεί να έρθει από τη Δυτική Αφρική στην Ευρώπη αναζητώντας ένα καλύτερο ε, οικονομικό μέλλον. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι σύνθετη η παρούσα εικόνα της μετανάστευσης και έχει πολλές αιτίες. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διευρύνουμε το πλαίσιο αναφοράς και να ελέγξουμε το σύνολο φάσμα των μεταναστευτικών φαινομένων που προκαλούνται από την αστάθεια. Αν δει κανείς τα στοιχεία που υπάρχουν, θα βρει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, μελέτες που κυρίως όμως ε, αποδίδουν τα πράγματα στην φτώχεια, στο χωμηλό ΑΕΠ, στην άνηση κατανομή του εισοδήματος, υψηλή ε, ανεργία, και προβλήματα περιβαλλοντικά. Ένα δεύτερο σύνολο αιτιών είναι η εθνοκάθαρση, οι πόλεμοι, οι συγκρούσεις. Το τρίτο είναι οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διακρίσεις, κακή διακυβέρνηση γενικότερα. Και τέλος θα μπορούσαμε επίσης να δούμε και τις φυσικές καταστροφές, είτε είναι ανθρωπογενείς, είτε είναι φυσικές όπως πλημμύρες, σεισμοί, ξηρασίες λοιπά. Λοιπόν, όταν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τις βασικές αιτίες της μετανάστευσης, θα πρέπει να ελέγξουμε τις πηγές αυτής της αστάθειας. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι υπεύθυνε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά σε περιφερειακό επίπεδο, στην Ασία, στην Αφρική κτλ να αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές ροές και τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν από τη χώρα τους είτε για πολιτικούς είτε οικονομικούς λόγους ε, δεν ε, έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, προσφεύγουν σε περιφερειακά κέντρα οικονομικής ανάπτυξης ή σε κέντρα θα έλεγα προσφύγων που τους παρέχουν μια κάποια προστασία. Τώρα, η πολιτική της μετανάστευσης μετά την Λισαβόνα είναι κοινή πολιτική, νεοπαγής πολιτική θα έλεγα, η οποία βοηθά να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά το θέμα της μετανάστευσης από τον πρώτο πυλώνα ε, σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, δεύτερος πυλώνας για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης όπου είναι εφικτή, και ε, τρίτος πυλώνας είναι η ενίσχυση και βελτίωση ε, των συνθήκων υποδοχής και να συνεισφέρουμε επίσης και στην ανάπτυξη ε, των χωρών προέλευσης, των μεταναστευτικών κυμάτων. Όπως είπα είναι το σημείο εκκίνησης αυτό, πρέπει να δούμε πέρα από την πολιτική μετανάστευσης, πρέπει να δούμε ας πούμε την εμπορική μας πολιτική η οποία θα πρέπει να έχει σαν στόχο την διασφάλιση θέσεων απασχόλησης στις χώρες προέλευσης, πρέπει να βελτιώσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης των προϊόντων από τις χώρες προέλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βοηθήσουμε να αναπτυχθούν τα εμπορικά περιφερειακά συστήματα που θα βελτιώσουν τον, την εμπορική δραστηριότητα νότου-νότου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για ό,τι συζητάμε σήμερα εδώ. Πρέπει να εξετάσουμε επίσης ε, και την πολιτική πρόληψη συγκρούσεων, να αποφύγουμε καταστάσεις απαράδεκτες, ε, να προχωρούμε σε διαιτησίες, να ενισχύουμε τα μέτρα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε χώρες με προβλήματα, να ελέγχουμε και να βοηθάμε τη σωστή ε, διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών να βοηθάμε στην κατάρτιση της αστυνομίας, της δικαστικής εξουσίας, όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Και φυσικά υπάρχει το θέμα της πρόσβασης στα τρόφιμα, στο καθαρό νερό, έτσι θα αποτραπούν μεταναστευτικές ροές οι οποίες οφείλονται σε αδυναμία επιβίωσης ουσιαστικά στις χώρες προέλευσης. Νομίζω ότι έτσι μόνο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις μετακινήσεις πληθυσμών ακόμα και στο εσωτερικό των χωρών από τις περιφέρειες στις μεγάλες πόλεις γιατί από τις μεγάλες πόλεις ξεκινούν τα μεγάλα μεταναστευτικά φαινόμενα. Πρέπει να δούμε επίσης και τις αρνητικές συνέπειες που προκαλούν μετανάστευση της κλιματολογικής αλλίωσης του πλανήτη ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φιλετικών δικαιωμάτων είναι πολλές φορές αιτία μεταναστευτικών πιέσεων. Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Βλέποντας τα όλα αυτά συνολικά είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί ορισμένα πολιτικά κόμματα που ασχολούνται ειδικά με την πίεση της μετανάστευσης ταυτόχρονα ασκούν κριτική στην αναπτυξιακή πολιτική. Αν θέλει να αντιμετωπίσει κανείς τις αιτίες της μετανάστευσης δεν μπορεί να αγνοήσει την αναπτυξιακή συνεργασία. Αν θέλει να αντιμετωπίσει την αστάθεια μπορεί να το κάνει αυτό αλλά πληρώνοντας το τίμημα. Πρέπει δηλαδή να ε, στηρίξει την ανάπτυξη και να βοηθήσει την αναπτυξιακή συνεργασία το τελικό θέμα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. <coughs> Είπαμε ότι έχουμε αρκετές πολιτικές, έχουμε πολλά μέσα στη διάθεσή μας και οικονομικά, εφόσον στοχεύουμε καλά την οικονομική μας παρέμβαση. Έχουμε γεωγραφικά μέσα παρέμβασης, θεματολογικά μέσα, επενδυτικά μέσα, Υπάρχουν και σφαιρικότερα μέσα για την σταθεροποίηση περιοχών, για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηματοδοτικά μέσα και τα μέσα που παρέχει και πά. Μπορούμε να πούμε ότι όλα τα οικονομικά μέσα για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά με την αντιμετώπιση της πραγματικής αιτίας της μετανάστευσης. Καθένα από αυτά τα μέσα βέβαια έχει κάποια κυρίαρχα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν στοχεύουν άμεσα στην μετανάστευση ή σε αυτούς που έρχονται και ζητούν άσυλο. Παρόλα αυτά όμως αντιμετωπίζουν άμεσα ή έμεσα και τις αιτίες της γενεσιουργίας της μετανάστευσης και της μεταναστευτικής πίεσης. Τέλος, ένα θέμα το οποίο μπορεί να επανέλθει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αν τα μέσα αυτά μπορούν να είναι πιο στοχευμένα στα πλαίσια της μείωσης των μεταναστευτικών ροών που προκαλούνται από περιφερειακές αστάθειες. Αυτό ίσως δεν είναι κάτι το απαραίτητο. Με ποια έννοια. Στόχος των μέσων αυτών είναι η μείωση της αστάθειας, είτε περιφερειακής, είτε πολιτικής, είτε οικονομικής. Εάν τα μέσα αυτά πετύχουν τους στόχους τους, τότε οι μεταναστευτικές ροές ε, θα ε, μειωθούν. Οι αυτές που προκαλούνται από την αστάθεια που έλεγα. Λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι εφόσον υπάρξει αποτελεσματική αναπτυξιακή βοήθεια, οι μεταναστευτικές ροές που οφείλονται στην έλλειψη ανάπτυξης θα μειωθούν. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τη συνεκτικότητα των πολιτικών μας, αλλά δεν υπάρχει ανάγκη νομίζω να υπάρξουν συγκεκριμένες πολιτικές που να στοχεύουν αποκλειστικά την μετανάστευση. Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα και αφού τα αναγνωρίζουμε μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και έτσι θα βοηθήσουμε να κατανοηθεί το πρόβλημα από όλους. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπρινέ. Καλημέρα σας. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρατού και τον κύριο Προβέρα για την ε, ε, πρόσκλησή μου να συμμετάσχω στην ακρόαση αυτή. Σήμερα θα σας κάνω μια παρουσίαση των ε, κατά πόσον είναι σημαντικό το πρόβλημα της μεταμνάστευσης σε σχέση με τις χώρες ε, που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στην Ευρώπη. Καταρχήν θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας δώσω κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που εξηγούν τη σημασία των προβλημάτων αυτών στις σχέσει με το Μαγκρέπ και κατόπιν θα σας δώσω κάποιες εξήγησεις πάνω στις λύσεις που προσπαθούμε να εγκαθιδρύσουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις πολιτικές μας. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εξηγούν τη σημασία της ε, μετανάστευση από το Μαγκρέπ το ένα είναι ότι είναι γειτονικέ χώρε κοντά στην Ευρώπη, γεωγραφική, ε, γεωγραφικά η απόσταση είναι πολύ μικρή και αυτό οδηγεί στο να περνάνε από εκεί και άλλα κύματα μεταναστευτικά που έρχονται από την Αφρική και από την Ασία και περνάνε ή από την Λιβύη προς τη Μάλτα ή από το Γιβραλτάρα χώρες δηλαδή διαμετακόμισης των, ε, της ε, μετανάστευσης αυτής. Από τις ίδιες τις χώρες αυτές βέβαια υπάρχει και ένα έντονο μεταναστευτικό ε, κύμα υπολογίζεται ότι 5 εκατομμύριο είναι οι οι προερχόμενα το Μαγκρέ που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το Μαρόκο βέβαια είναι ακόμα μεγαλύτερα τα ποσοστά αυτά. Το δέκατο, το δέκατο του πληθυσμού του Μαρόκου ζουν περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα οδηγεί σε προβλήματα ανθρώπινα, πολιτιστικά, ανισορροπίες μεταξύ των διαφόρων ε, κοινωνών αυτών σημαντικά, σημαντικές και αυτό που είναι σημαντικό είναι η σχέση που έχουν επίσης αυτές οι ε, συνοικίες αν θέλετε ε, Μαγρεμπίνων στην Ευρώπη με την χώρα που είναι Υπάρχει ένας σημαντικός δυναμισμός και μια φυσική πίεση δημογραφική. Υπολογίζεται ότι ότι ο πληθυσμός των τριών κεντρικών ε, χωρών του Μακρέπ θα αυξηθεί κατά πάνω από 25 εκατομμύρια μέχρι το 2050, θα περάσει λέει δηλαδή από 75 στα 105 εκατομμύρια μέχρι το 2050 αυτό δεν θα ήταν βέβαια πρόβλημα εάν στις χώρες αυτές υπήρχαν αρκετές δυνατότητες απασχόλησης. Όμως ένα μεγάλο πρόβλημα του Μαγκρέπ και γενικά του αραβικού κόσμου αυτή τη στιγμή είναι η αδυναμία να δημιουργηθούν επαρκείς θέσεις απασχόλησης ή να απασχολήσουν όλους αυτούς τους νέους που θα περάσουν στην αγορά εργασίας. Υπολογίζεται ότι για την Αλγερία, Μαρόκο και την Ισία μέχρι το 2020, σε 10 χρόνια δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργήσουν 5 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης και να απορροφήσουν μόνο και μόνο τους νέους, να σταθεροποιήσουν δηλαδή τα ποσοστά ανεργίας που είναι σήμερα αρκετά υψηλά. Οι χώρες αυτές θα πρέπει να δημιουργήσουν δηλαδή θέσεις απασχόλησης με μεγαλύτερη ταχύτητα, αυξάνοντας ταχύτητα αυτή κατά 50%. Υπάρχει λοιπόν εδώ το πρόβλημα αυτό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ενδεχόμενης βέβαια ε, οικονομικής αστάθειας. Γιατί δεν θα υπάρχουν προοπτικές εργασίες ε, στην χώρε στις χώρες αυτές. Δεν μπορούν να δημιουργηθούν εκεί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η απόσταση εισοδημάτων μεταξύ του Μαγκρέφ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 1 προ 10 μεταξύ των τριών χωρών του mm. Κεντρικού Μακρέπ και της Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η μεγαλύτερη απόσταση ε, μεταξύ δύο γειτονικών χωρών. παραδείγματο χάρη ε, μεταξύ ε, Μεξικού και ΙΠΑ είναι 1 προ 4, 1 προ 5. Η διαφορά λοιπόν εισοδήματο ε, μεταξύ Μακρέπ και Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνει ακόμα περισσότερο την πίεση που ασχείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγιναν κάποιες μελέτες και θεωρήθηκε ότι πάνω από το 50% των νέων στο Μαγκρέπ θέλαν να μεταναστεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε μια πρόσπαση ανάλυση ένα, ε, ε, ε, από ένα ίδρυμα στο το Λοφίν που είπε ότι το 37% ε, εκείνο που ερωτήθηκαν πού θα θέλαν να πάνε για να ξανακάνουν μια καινούρια ζωή, το 37% λέω ήθελαν να πάνε στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν σημαντική πίεση. Όταν το γνωρίζουμε αυτό, ποιες είναι περίπου οι λύσεις που έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε ή θα πρέπει να εφαρμόσουμε στο μέλλον. Όπως είπε και ο συνάδελφος, το κεντρικό σημείο ήταν να έχουμε μια σφαιρική αντιμετώπιση της μετανάστευσης, να υπάρχει δηλαδή μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα πρέπει να εξετάζει αυτά τα προβλήματα της μετανάστευσης σε όλες τις πτυχές. Απασχόληση, οικονομική, εμπορική, ανάπτυξη, ακόμα και η πολιτική που ασχολείται με αυτή καθ' την μετανάστευση ή την ε, φύλαξη των συνόρων. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα με τις χώρες που το επιθυμούν, αναπτύσσει μία ατζέντα οικονομική που αυξάνει τις ευκαιρίες στις οικονομικές στις χώρες του Μαγκρέπ. Στο Μαρόκο και τη, την Ισία έχουμε στα πλαίσια της πολιτικής γυτνίασης τα πιο αναπτυγμένα σχέδια Και αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί ιδίω όσον αφορά την ανάπτυξη των πολιτικών απασχόληση. Για τι χώρε αυτέ η πολιτική απασχόληση δεν είναι επαρκώ προσανατολισμένη προ τη δημιουργία απασχόληση καλή και παραγωγική. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια. Πιο γενικά, όσον αφορά τη μετανάστευση, θα πρέπει να υπάρχει μια πιο συνεπής προσέγγιση, να υπάρχει δηλαδή μια εταιρική σχέση με τις χώρες του Μαγκρέπ που άπτεται των διαφόρων ε, πτυχών της σφαιρικής προσέγγισης. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό μέσα πλαίσια της ατζέντας συνεργασίας που ε, υπογράψαμε τη Λιβύη, προσπαθώντας να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Λιβύης και των χωρών νότια της Σαχάρας, από τους οποίους προέρχεται η μετανάστευση, ούτω ώστε να μπορέσουμε έτσι να ενδυναμώσουμε τις οικονομικές δυνατότητες της Λιβύης προς όφελος των χωρών από τους οποίες προέρχονται οι μετανάστες αυτές και ταυτόχρονα έλεγχος και διαχείριση της νόμιμης ε, μετανάστευσης στη Λιβύη μέσα διαχείρισης της μετανάστευσης και προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε όλα αυτά που αφορούν την προστασία των μεταναστών που χρειάζονται μια διεθνή προστασία. Είναι πραγματικό πρόβλημα αυτό των δικαιωμάτων των προσφύγων παραδείγματο χάρη, γιατί αυτές οι χώρε του Μαγκρέπ τώρα όσο πάει και περισσότερο γίνονται χώρε προορισμού τη μετανάστευση ή τουλάχιστον διαμετακόμιση τη μετανάστευση. Και θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι επίσης σημαντικό όσον αφορά την διαχείριση του ελέγχου των συνόρων, γιατί όπως σας είπα αυτές οι χώρες του Μαγκρέπ υπόκεινται στην άτακτη αυτή η μετανάστευση που τους παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα. Αυτό ισχύει για την Λιβύη αλλά και άλλες χώρες όπως το Μαρόκο, την Αλγερία που πλήττονται από αυτό το πρόβλημα. Το παράδειγμα της Λιβύης είναι ενδιαφέρον γιατί για πρώτη φορά μπορέσαμε να αναπτύξουμε μια δέσμη συνεκτική και σφαιρική για τον τομέα της ε, μετανάστευσης. Δυστυχώς ε, δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα με τις άλλες χώρες. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπημένη εταιρική σχέση, διαφοροποιημένη που άπτεται όλων των προβλημάτων. Μέχρι στιγμής τονίστηκε ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλειας, ιδίω όσον αφορά τις συμφωνίες επαναπατρισμού ή επανιστοχής, mobilité euh, n'a pas été euh, suffisamment développée. Και αυτό δικαιολογεί, νομίζω, εξηγεί τουλάχιστον την, ε, ε, το δισταγμό ορισμένων χωρών. Θα πρέπει πάντως να αναπτύξουμε με το Μαγκρέπ μια πιο φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της μετανάστευσης και θα σας δώσω εδώ δύο στοιχεία προσκέψη. Όσα αφορά την Τριμερή συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης, των χωρών του Μαγκρέφ και των χωρών νότια της Ζαχάρας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μέσα στα μέσα που έχουμε θα πρέπει να αναπτύξουμε αυτή την πτυχή της συνεργασίας, της τριμερούς συνεργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και τελευταίο, δεν θα πρέπει να ε, περιορίσουμε την προσοχή μας σε προβλήματα της ασφάλειας μόνο, αλλά να εξετάσουμε σφαιρικά όλα τα προβλήματα της μανάστευσης και να αναπτύξουμε ένα πιο φιλόδοξο ε, σχέδιο πολιτικής για την κινητικότητα των ατόμων και να έχουμε ε, μια εταιρική σχέση στην οποία όλοι κερδίζουν με τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Stavo scrivendo e quindi ritardo un poco nel, nel dare θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πάτσε. Ladies Κυρίε και κύριοι, κυρία Προβέρα, κύριε Κρετού, είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σήμερα εδώ. Μιλάμε για την μετανάστευση, ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ένα θέμα πάνω στο οποίο εργάζομαι και εγώ θέλω να αναφερθώ πάνω στην αναγκαστική μετανάστευση και μια σφαιρική προσέγγιση. και τη διαχείριση της ε, μετανάστευσης μέσα στα πλαίσια του κράτους δικαίου. Θα μιλήσουμε επίσης για ορισμένες προκλήσεις του σφαιρικού αυτού φαινομένου. Αρχίζοντα με το πρώτο σημείο, μπορούμε να πούμε ότι η διάκριση ε, υποχρεωτικής ε, μετανάστευσης και μη αναγκαστικής ε, δεν είναι πια τόσο έντονη. Ο συνάδελφος Ρούδος στην αρχή αναφέρθηκε στον δυναμισμό που υπάρχει πίσω από το φαινόμενο της μετανάστευσης. Θα πρέπει να το ορίσουμε σαν ένα φαινόμενο, ένα γεγονός αν θέλετε, δεν είναι μόνο πρόβλημα. Και θα πρέπει να εξετάσουμε την μετανάστευση πολύ πιο σφαιρικά. ξέρουμε ότι η διεθνής μετανάστευση συμπεριλαμβάνει και τους πρόσφυγες και άλλα άτομα που δεν ε, μπορούν να μείνουν στις πατρίδες τους. Αν κοιτάξουμε την αναγκαστική αυτή μετανάστευση μπορούμε αμέσως να μιλήσουμε για πρόσφυγες. Ε, Σύμβαση 1951. Αλλά χρησιμοποιούμε και τον όρο των εκτοπιστέντων. δηλαδή άτομα τα οποία δεν έχουν αναγκαστικά εκτεθεί σε διώτες αλλά που αναγκάζονται να φύγουν από εκεί που κατοικούν για διάφορους λόγους καταστροφών κλπ. Αυτό συμπεριλαμβάνει και εκείνους που μένουν μέσα στις χώρες τους, στα σύνορά τους ή που έχουν περάσει τα σύνορα. Και έχουμε διάφορες, διάφορους φεούς εδώ. Παραδείγματο χάρη είναι μετανάστευση που οφείλεται σε περιβαλλοντικού λόγου. Περιβαλλοντική αυτό λόγο θα μπορεί πραγματικά να είναι και αυτή ένα λόγο μετανάστευση. Περιβαλλοντική αυτή μετανάστευση μπορεί να είναι εσωτερική ή και διεθνή. Και μπορούν πολλοί επίση να εκτοπιστούν για λόγο καταστροφών φυσικών ή μη φυσικών. και αυτό μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. Η, ε, ε, επίσης αυτή η μετανάστευση όταν αυξηθεί μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ε, περιβαλλοντικά προβλήματα. Έχει αυξηθεί πια το μέγεθος της μετανάστευσης γιατί βλέπουμε από το 98 στη 2007 2,2 δισεκατομμύρια ατόμων πλήγησαν από καταστροφές, ενώ στην προηγούμενη δεκαετία ήταν 1,8 δις. Υπάρχει λοιπόν πάρα πολύ σημαντική αύξηση. Αν κοιτάξουμε από την άλλη πλευρά βέβαια του φάσματος, υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μεταναστεύουν χωρίς να υποχρεούνται από κάποιους εξωτερικούς παράγοντας. Εθελοντικά κύματα δηλαδή. 214 εκατομμύρια ατόμων ε, έχει εκτιμηθεί ότι είναι αυτοί οι διεθνείς μετανάστες και οι περισσότεροι αυτοί από αυτούς είναι μεταναστές εργαζόμενοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους. Η διάκριση λοιπόν στην οποία αναφέρεται στο, στην αρχή μεταξύ της καταστικής και της εθελοντικής μετανάστευσης δεν είναι πια τόσο αυστηρή. Γιατί η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε μια χώρα και να αναγκάσει τους κατοίκους εκεί να ζητήσουν μια καλύτερη τύχη αλλού. Είναι δύσκολο να ε, διακρίνουμε μεταξύ των ομάδων. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να κάνουμε κάποιες διακρίσεις γιατί υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες που ισχύουν διαφορετικές ομάδες. Υπάρχουν βέβαια και κοινά σημεία. Είναι άνθρωποι όλοι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανθρωπιστική, η ανθρώπινη πλευρά, αν θέλετε. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, όταν μιλάμε γενικά για τη μετανάστευση και πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διάφορες κατηγορίες ε, ατόμων που μεταναστεύονται, ότι θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και εκεί, παραδείγματος χάρη, εκμετάλλευση. Πρόσφατη περίπτωση αυτές οι χιλιάδες οι, χιλιάδες ε, <clears throat> μετανάστες που ε, βρέθηκαν να ζουν χωρίς νερό, χωρίς ηλεκτρισμό σε μία από τις χώρες μέλη. Άνθρωποι που είχαν έρθει στην Ευρώπη γιατί τους είχαν υποσχεθεί ε, δουλειά επίσημη και όταν έφτασαν εδώ η δουλειά που, που βρήκανε ήταν τελείως ανεπίσημη στη μαύρη και κάτω από πάρα πολύ κακές προϋποθέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα δεδομένο ζωής ε, η μετανάστευση και ο ρόλος που μπορεί να παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά η Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Στο δεύτερο σημείο της συζήτησή μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα σετ προτύπων για να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είπαμε ότι μιλάμε για ανθρώπους, ε, για ανθρώπους που έχουν δικαιώματα. Και υπάρχουν διάφοροι νόμοι διεθνείς ή και εθνικοί που εφαρμόζονται για τους ανθρώπους αυτούς δεν πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε την επέτειο πριν, που πριν από 20 χρόνια ε, υιοθετήθηκε μια σύμβαση για τα δικαιώματα των μεταναστών αυτών. Πολλές αρχές ε, υπάρχουν, παραδείγματος ανθρωπιστική αντιμετώπιση, ε, συνεργασία, μη παρέμβαση, πρόληψη, ε, ετοιμότητα πολλές αρχές οι οποίες εφαρμόζονται και στην περίπτωση ε, καταστροφών. Είναι ουσιαστικό, όπως είπαμε, το θέμα να εξετάσουμε τις ε, καταστροφές. Αυτό είναι το κέριο σημείο για την προστασία μετά την καταστροφή και κατά διάρκεια της ανοικοδόμησης στο μέλλον but the protection of those involved in migration, the right to humanitarian assistance. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί βέβαια να αποχωριστεί από την υποχρέωση να προληφθούν οι καταστάσεις οι οποίες οδηγούν σε βία, οι οποίες οδηγούν σε αστάθεια. Και επίσης η κατεπίγουσα βοήθεια έχει σαν στόχο ακριβώς την προστασία της ζωής. θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πληθυσμών αυτών θα πρέπει να παραμείνει εξίσου ισχυρή σε όλα τα στάδια. Ένα κράτος έχει βέβαια την υποχρέωση να προστατεύσει όλους τους πολίτες. Το αναγνωρίζουμε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι κάποιοι διεθνείς ε, δράσεις μπορούν να βοηθήσουν μια χώρα σε αυτή την, ε, σε αυτή την προσπάθεια της προστασίας. Να μην υπάρχουν, ας παραδείγματος χάρη, το εμπόριο των ανθρώπων αυτών, να τους δίνουν τη δυνατότητα μεταφορά, ε, μεταφορικών μέσων σε περίπτωση διαμαχών. Να μπορεί δηλαδή αυτό το κύμα να ελέγχεται με ανθρώπινο τρόπο. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ σημαντικός και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα περισσότερο από το παρελθόν γιατί τώρα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε πολύ υψηλό, υψηλή σημασία βάσει τη συνθήκης της Λισαβόνα. Όταν ε, περάσουμε στο τρίτο σημείο που μιλάμε για τη σχέση μεταξύ των περιβαλλοντικών καταστροφών ε, και των ε, μετασταυτικών ροών, θα πρέπει να περάσουμε νομίζω από την αντίδραση μονάχα σε καταστροφές σε μια πιο συλλογική, προληπτική, έγκαιρη παρέμβαση είδαμε πολλά στο παρελθόν και καταλήξαμε σε καλά διδάγματα με τη συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους όσον αφορά την κατεπίγουσα βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών ή την ε, προσαρμογές του κλίματος ε, λόγω της μετανάστευσης Μιλήσαμε προηγουμένω για το Μάγκρεπ και θα ήθελα να αναφερθώ σε συγκεκριμένε θέσει όσον αφορά ακριβώ αυτέ τι αλλαγέ ε, θεματολογικέ ε, λόγω τη μετανάστευση στην Αίγυπτο. Εκεί υποστηρίζουμε την Αιγυπτιακή κυβέρνηση να ε, ενισχύσει τι δραστηριότητε για να την αύξηση του, της στάθμης του Νείλου γιατί εάν αυξηθεί η στάθμη της θάλασσας θα μπορέσει να εκτοπίσει εκατομμύρια ατόμων. Και προσπαθούμε να δούμε ποιες θα είναι πραγματικά οι επιπτώσεις στη μετανάστευση αν υπάρχει η αύξηση της στάθμης αυτής και πώς θα μπορέσουμε να αντιταχθούμε και να αντιδράσουμε τώρα. Θα μπορούσε παραδείγματο χάρη να γίνει κάτι για να αυξηθούν οι δυνατότητες των πληθυσμών που ζουν σε περιοχές που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη του σχετικά με τη θάλασσα. Το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία ή για την Κολομβία. Υπάρχουν παντού τέτοιες δυνατότητες που θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ανθρώπους που απειλούνται από κάποια φυσική καταστροφή στο μέλλον. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Και εδώ σήμερα συζητάμε και ταυτόχρονα στο Τζιμπουτί υπάρχει ακριβώς μια, ένα συνέδριο για να δούνε πώς θα μπορούν να αντιμετωπίσουν την περίπτωση στην οποία υπάρχει αυτή η μετανάστευση λόγω ε, καταστροφών στο Τζιμπουτί και στη γύρω περιοχή η άδακτη αυτή μετανάστευση είναι σε πολύ υψηλούς ρυθμούς. Τι μπορούμε να κάνουμε, εμεί τι μέσα έχουμε για να αντιδράσουμε αποτελεσματικά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, το τελευταίο είναι αυτό που θέλω να αναφέρω. Θα πρέπει να υπάρχει καταρχήν χρηματοδότηση για την φάση της ε, έγκαιρης ε, αντιμετώπισης είπα ότι πολλές φορές είναι εύκολο να έχει κανένας την περίπτωση της, ε, της καταστροφής, ε, στη στιγμή της καταστροφής, αλλά μετά για την ενοικοδόμηση είναι πολύ δύσκολο. Πολλές φορές τα χρήματα φτάνουν όταν έχει ξεκινήσει η φάση της ε, ανοικοδόμησης και αυτό δεν επιτρέπει να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις που έχουν συλλέξει κατά τη διάρκεια της ε, επίγουσας κατάστασης. Τονίζεται επίσης ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούμε χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη της συνοχής, γιατί δημιουργείται απλώς μία εξάρτηση. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει η συνοχή και να μην υπάρχει κενό μεταξύ της κατεπίγουσας κατάστασης και της ε, ε, φάσης ανοικοδόμησης. Προσβλέπω τη συζήτηση και στα σχόλιά σας. Σας ευχαριστώ. Η τελευταία παρέμβαση είναι του κυρίου Μόρα Μπεναβέντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου στείλετε ε, και σας κυρία Κρέτσου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί μου δίνετε ιδιαίτερη χαρά και μου κάνετε την τιμή να μιλήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ συμφωνούμε ότι οποιαδήποτε μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να έχει και μία συνιστόσα εξωτερικής πολιτικής. Η έλεγχη στα σύνορα είναι μάλλον απαραίτητη και καλή, αλλά δεν δίνεται να, δεν να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ουρές μόνο με τον έλεγχο των συνόρων και εσωτερικές πολιτικές όπως πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγεία είναι σημαντικές αλλά δεν μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα. Είναι σημαντικές πολιτικές αλλά και πάλι δεν αλλάζουν τις τάσεις στις χώρες προέλευσης. Όταν λοιπόν χρειαζόμαστε μία εξωτερική πολιτική, θα πρέπει να απαντήσουμε σε τρεις ερωτήσεις, για να δούμε πώς θα την χαράξουμε και πώς θα την εφαρμόσουμε. Πρώτο ερώτημα είναι, τι, πώς αντιμετωπίζουμε την ε, μετανάστευση υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής. Δεύτερον, ποιες είναι οι διασυνδέσεις ε, μετανάστευσης και εξωτερικής πολιτικής. Και τρίτον, πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξωτερική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τα μεταναστευτικά θέματα. Πρώτη ερώτηση. Πώς μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μετανάστευση υπό το πρίσμα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση. Η εξωτερική πολιτική έχει στόχο την διαφύλαξη της σταθερότητας και της ασφάλειας, αφενός, αλλά και ε, την πρόθεση των ευρωπαϊκών συμφερόντων αφετέρου. Όταν λαμβάνουμε υπόψη ότι μαζικές μεταναστευτικές ουρές, κυρίως λάθρο μεταναστών, θεωρούνται ως απειλή στην σταθερότητα και την ασφάλεια, μπορούμε εύκολα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι χρειαζόμαστε την εξωτερική πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι με βάση τον τίτλο «Μεταναστευτικές ώρες που προκύπτουν από την αστάθεια» εγώ θα αναφέρω με στη διάρκεια της ομιλίας μου περισσότερο στην α, λαθρομετανάστευση γιατί η ελεγχόμενη και νόμιμη μετανάστευση είναι σημαντικό εργαλείο σίγουρα εξωτερικής πολιτικής. Για παράδειγμα, η πολιτική που ακολουθούν οι Ηνωμένε Πολιτείες Να προσελκύσουν τους εκλεκτούς, τους ε, φιέστερους από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Και παρόλο που έχουν αυστηρά μέτρα εξωτερική πολιτική, αυτή η πολιτική του για να προσελκύσουν του καλύτερου, του πιο εκλεκτού, είναι ε, σημαντική. Έχουμε και άλλα εργαλεία, soft policy, αλλά εδώ δεν μιλούμε για την νόμιμη και ελεγχόμενη μετανάστευση, εδώ μιλούμε για την λάθρο μετανάστευση, την ανεξέλεκτη. Και αυτές οι μαζικές μεταναστευτικές ροές πολλές φορές δημιουργούν αστάθεια, γι' αυτό χρειαζόμαστε την εξωτερική πολιτική για να την αντιμετωπίσουμε. Θα ήθελα όμως να κάνω εδώ δύο διευκρινήσεις, γιατί η εξωτερική πολιτική που εφαρμόζουμε θα μεταβάλλεται και θα διαμορφώνεται με διαφορετικό τρόπο. Η ασφάλεια και η σταθερότητα εκλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το γεωγραφικό αλλά και το χρονικό πλαίσιο. Σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία η μετανάστευση γίνεται αποδεκτή πολύ πιο εύκολα από ότι σε πιο ομοιόμορφες και ομοιογενείς κοινωνίες. Κάτι που κάποια χρονική στιγμή θεωρείται απειλή, σε άλλη χρονική στιγμή δεν θεωρείται κατά ανάγκη απειλή. Όλα αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη ότι έχει σημασία το γεωγραφικό και το χρονικό πλαίσιο για την εφαρμογή δεδομένη εξωτερική πολιτική. Επίση, οι απειλέ, οι πραγματικέ απειλέ ε, και πάλι γίνονται αντιληπτέ με διαφορετικό τρόπο. Η χάραξη όμως και η διαμόρφωση της πολιτικής θα πρέπει να γίνει με βάση τις ε, πιθανέ απειλέ αυτές που αντιλαμβανόμαστε ω απειλές. Αυτό ζητάει η κοινή γνώμη. Είχαμε πρόσφατο παράδειγμα πάλι από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ήταν διαφορετική η αντίληψη της κοινωνίας της Αριζόνας για την μετανάστευση από το Μεξικό σε σχέση με την αντίδραση των πολιτιών Σικάγο και Ιλινόης, για παράδειγμα. Λες και οι πολιτείες αυτές ανήκαν σε διαφορετικές χώρες. Και η χάραξη εξωτερικής πολιτικής προς το Μεξικό, για παράδειγμα, εκ μέρους των Πολιτειών, θα πρέπει να γίνει υπό το πρίσμα της α, θεωρούμενης απειλής, όχι κατά ανάγκη της πραγματικής απειλής. Οπότε, υπάρχει το θέμα της διασύνδεσης ε, ως προς την αστάθεια και την ε, ασφάλεια και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Έρχομαι στο δεύτερο ερώτημα, συσχετισμός μετανάστευσης και εξωτερικής πολιτικής. Η μετανάστευση είναι κυρίως εσωτερική πολιτική. Στις χώρες σας λαμβάνετε διαφορετικά μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, για παράδειγμα έλεγχη στα σύνορα κτλ. Αλλά οι πολιτικές αυτές έχουν και εξωτερικές επιπτώσεις και στην περίπτωση της, μεταναστευτικής, της μετανάστευσης αυτές οι εξωτερικές συνέπειες μπορεί να είναι τεράστιες. Οπότε είναι σαφής ο συσχετισμός. Χρειαζόμαστε την εξωτερική πολιτική για να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες των εσωτερικών μας πολιτικών για τη μετανάστευση. Όπως είπα, η μετανάστευση μπορεί να είναι μαζική και μεγάλη. Μπορεί να δημιουργηθεί ένας τεράστιο διμερές πρόβλημα με τις χώρες προέλευσης, με τις χώρες διέλευσης, ακόμη και με την ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκουν αυτές οι χώρες. Και πολλές φορές στο παρελθόν είδαμε πόσο γρήγορα μπορεί να επιδεινωθεί η κατάσταση και οι σχέσεις μεταξύ της χώρας προέλευσης και της χώρας ε, προορισμού υποδοχής. Και υπάρχουν πολλές ε, πιθανές πηγές και αιτίε έντασης και σύγκρουσης μεταξύ των δύο χωρών προέλευσης και προορισμού. Η πρώτη γνωστή για μας κατάσταση είναι όταν εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούμε τις χώρες προέλευσης επειδή δεν λαμβάνουν, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, αρκετές δράσεις για να αποτρέψουν αυτές τις μαζικές μεταναστευτικές ροές. Υπάρχει όμως και άλλη όψη του νομίσματος. Οι χώρες προέλευσης ε, κάνουν χρήση και κατάχρηση μερικές φορές αυτής της κατάστασης για να διεκδικήσουν ε, οικονομικά, εμπορικά πλεονεκτήματα ή προνόμια ή και για λόγους στρατηγικής. Και πολλές φορές, παραλαμβάνω, γίναμε μάρτυρες της ταχής επιδείνωσης αυτής της κατάστασης. Γι' αυτό και θα πρέπει να αντιδράσουμε χρησιμοποιώντας την εξωτερική πολιτική για να αποφύγουμε τον εκτροχιασμό. Υπάρχει όμως και μια άλλη πηγή πιθανής σύγκρουσης και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε εμείς τι κάνουμε. Ποια είναι η συμπεριφορά τη κυβέρνηση ή ποια είναι η συμπεριφορά των κοινωνιών μας απέναντι στους μετανάστες. Και δεν μιλώ μόνο για τη γενική αντίληψη και τη, μια ξενοφοβία. Μιλώ για συγκεκριμένα πράγματα. Πρόσβαση στην παιδεία, πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Όταν λοιπόν ε, και η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται και πάλι υπάρχει πρόβλημα. Ένα παράδειγμα είναι οι μουσουλμάνοι μετανάστες στην Ευρώπη. Σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα αντιμετωπίζει πολλές φορές ε, διαδηλώσεις μπροστά σε ε, πρεσβείες μουσουλμανικών χωρών. Ξέρετε τι εννοώ. Και αυτό επηρεάζει την αντίληψη τη κοινωνία. Αυτό είναι θέμα εσωτερική πολιτική που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Υπάρχει και κοινωνική πτυχή. Για να αντιμετωπιστεί όμω σωστά αυτή η κοινωνική εσωτερική πτυχή χρειαζόμαστε και μια εξωτερική πολιτική, μια εξωτερική πολιτική απέναντι στι χώρε προέλευση. Αλλιώ και πάλι ελοχεύει ο κίνδυνο τη επιδείνωση τη κατάσταση. Και τώρα ένα σύντομο σχόλιο για διαμετρικά αντίθετη κατάσταση. Μίλησα για τι ε, διεθνεί συνέπειε των εσωτερικών πολιτικών. μερικέ φορέ όμω. Ε, τα κριτήρια της εξωτερικής πολιτικής είναι κρίσιμα και με τον ένα τον άλλο τρόπο επηρεάζουν και το πόσο γίνονται αποδεκτές οι εσωτερικές πολιτικές μετανάστευσης. Για παράδειγμα, οι χώρες μέλη που δεν αντιμετώπισαν το κοσυφοπαίδιο και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους κοσοβάρους μετανάστες είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αλλιώς αντιμετωπίζουν λαθρομετανάστες μια χώρα που αναγνώρισαν και αλλιώ αντιμετωπίζουν μετανάστε μια χώρα που δεν έχουν αναγνωρίσει. Και έρχομαι στο τρίτο ερώτημα. Πώ χρησιμοποιούμε την εξωτερική πολιτική για να διαχειριστούμε τη μετανάστευση. Όταν έχουμε μια κατάσταση όπου πιστεύουμε ότι θα απειληθούν η σταθερότητα και η ασφάλειά μας, σκεφτόμαστε αμέσως την αποτροπή. Αλλά η αποτροπή σε θέματα μετανάστευσης είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι όταν δεν χρησιμοποιούμε στις διεθνείς σχέσεις. Χρειάζεται αλλαγή της νοοτροπίας της συμπεριφοράς των κυβερνήσεων. Και εδώ έχουμε χιλιάδες ή εκατομμύρια ανθρώπους που ο καθένας για τους λόγους του και για τα συμφέροντά του έρχονται εδώ. Πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους, στη ζωή τους Οπότε είναι πολύ περίπλοκη η κατάσταση. Χρειαζόμαστε ό,τι εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μα, οποιοδήποτε μηχανισμό τη εξωτερική πολιτική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, ελεύθερο εμπόριο. Δεν έχει νόημα να, να τεράστια, επειδή τεράστια ποσά προς τις χώρες αυτές, ενώ με ένα μικρότερο, με ένα μικρότερο οικονομικό, με μικρότερη οικονομική επένδυση θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τις άμεσες επενδύσεις στις χώρες αυτές, με την βοήθεια την αναπτυξιακή, με την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Είναι ένα άλλο είδος εξωτερικής πολιτικής που θα πρέπει να επιδιώξουμε στις χώρες αυτές, πέραν της οικονομικής βοήθειας. Επίσης, διμερείς συμφωνίες με τις χώρες αυτές που δεν θα περιορίζονται στη μετανάστευση αλλά σε όλες τις πτυχές της προστασίας των μεταναστών ώστε να αποφύγουμε τη διάδοση αυτών των διμερών συγκρούσεων όταν ανακύπτουν ή περιφερειακές προσεγγίσεις. Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το Σαχέρ, για τη Σαχάρα, μάλλον την υποσαχάριο Αφρική. Η ε, ο συνάδελφος μίλησε για το Μαγκρέπ πριν. Το Σαχέλ είναι μια περιοχή όπου εξαιτίας της μακροχρόνιας ξηρασίας δημιουργήθηκαν τεράστιες μεταναστευτικές ροές από την περιοχή Σαχέλ. Η συνάδελφος εδώ έχει ένα βιβλίο για, την, για τις κλιματικές αλλαγές και με τη μετανάστευση. Αυτή ήταν ίσως η πρώτη οικολογική μετανάστευση. Αλλά ούτως ή άλλως ε, η μετανάστευση, οι αστάθειες χώρες αυτές είναι κάτι κοινό, γιατί μπορεί να μην είναι ε, χώρες ε, ταραξίες κατά ανάγκη, αλλά είναι σχεδόν χώρες στις οποίες επικρατεί χάος. Και μάλιστα έχουμε στοιχεία που μας δείχνουν ότι μόνο ένα στους έξι μετανάστες από την περιοχή Σαχέλ, Σαχέλ ήρθαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υπόλοιποι πέντε στους 6 έμειναν στην περιοχή. Χρειαζόμαστε μια περιεκτική προσέγγιση για την περιοχή Σαχέλ, όχι μόνο για την μετανάστευση, γιατί πέραν της μετανάστευσης ε, είχαμε και άλλα προβλήματα, τρομοκρατία, λαθρεμπόριο ναρκωτικών κτλ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια συνολική περιεκτική στρατηγική την επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μία όθηση προς την κατεύθυνση αυτή και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν χρήσιμη για την ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις γνώσεις που μας δώσατε, για την εμπειρία σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Η κυρία Λόχμπίλερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους εμπειρογνώμονες για τις αναλύσεις τους που ήταν πολύ εμπεριστατωμένες. Κύριε Μπρουνέ, είπατε ότι τρεις είναι οι πυλώνες της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ευρώπη. Έχουμε βέβαια και το σχετισμό εξωτερικής και μεταναστευτικής πολιτικής. Έχουμε βέβαια και την νόμιμη μετανάστευση. Ασχοληθήκατε κυρίως με την λάθρο μετανάστευση. Δεν μπορούμε να είμαστε αξιόπιστοι στην εξωτερική μας πολιτική αν δεν ασχοληθούμε και με το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Ο κύριος Μποναβέντε και ο κύριος Ρόζεμπορκ μίλησαν και για αναγκαστική μετανάστευση εξαιτία των κλιματικών αλλαγών. Αυτό το ανέφερε και η κυρία Πάτσε. Ο κύριος Ρόζεμπορκ μας είπε ότι 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάζονται να μεταναστεύσουν εξαιτίας των θεομηνιών. Και είναι διαφορετικές οι προβλέψεις για το ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των μεταναστών που έχουν επηρεαστεί από τις θεομηνίες. Έχει στοιχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση για το ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και θεομηνίες. Αναφέρθηκαν κάποια στοιχεία για την περιοχή του Μαγκρέπ. η Ελλάδα ζήτησε από τη Frontex, τον Οργανισμό Προστασίας των Συνόρων, να εξασφαλίσει τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, γιατί αν δεν είμαστε προσεκτικοί σε αυτόν τον έλεγχο θα έχουμε τεράστια ροή μεταναστευτική μεταναστών. Στην Τουρκία δεν ισχύει δίκαιο για το άσυλο. Επίσης στο Ιράν σε σχέση με το 2009 είχαμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών κατά 30%. Ιδιαίτερα ετούν τον άσυλο οι ανθρώπων που υπόκεινται σε πολιτική δίωξη στο Ιράν ή στην Τουρκία. Ο κύριος Παναβέντε μίλησε για την προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους. Γνωρίζετε όμως ότι κανένα κοινοτικό κράτος δεν έχει υπογράψει αυτή την συνθήκη ή τουλάχιστον δεν έχει, εφαρμόσει, και δεν έχει εφαρμόσει. Γιατί τα κράτη-μέλη, κατά τη γνώμη σας, δεν υπογράφουν αυτή τη συνθήκη για την προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους. Νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε πια μια νέα εντολή, ένα θέμα που συζητήσαμε στην Επιτροπή μας για την Frontex, τον Οργανισμό δηλαδή Προστασίας των Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υποβάλουμε μια σύσταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο που γίνεται η κατάρτιση, για τις αποστολές, για την αξιολόγηση αυτού του οργανισμού. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο, στην εντολή της Frontex και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να παρακολουθεί Frontex και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πολύ πιο αυστηρά. Η κυρία Κέλλερ από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε ο κύριος Μπρουνέ. Συμφωνώ και με τον κύριο Μπρουνέ και με τον κύριο Ρόζεμπορκ ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τη μετανάστευση όταν μιλούμε για ανάπτυξη. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά δεν υπάρχει στενή σχέση μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών διέλευσης και των μεταναστευτικών ροών. Θα πρέπει να εξελίψουμε τους όρους της συνθήκης της αστάθειας, τις αιτίες της αστάθειας δεν αρκεί να δίνουμε αναπτυξιακά κονδύλια στις χώρες διέλευσης. Δεν αρκεί αυτό για να σταματήσουμε τα αίτια της μετανάστευσης. Συμφωνώ όταν μιλούμε για τη μετανάστευση να λαμβάνουμε υπόψη και την αναπτυξιακή μας πολιτική, αλλά διαφωνώ με την χορήγηση αναπτυξιακών κονδυλίων για την εξασφάλιση των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που δυστυχώς ε, συμβαίνει αυτή τη στιγμή ελπίζω να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κονδύλια να φτάνουν στο σωστό προορισμό και να είναι αναπτυξιακά να χορηγούνται όντω για την ανάπτυξη. Ο κ. Δεμπρόκη αναφέρθηκε στο ελεύθερο εμπόριο που θα βοηθήσει την ανάπτυξη, θα αποκαταστήσει κάποια σταθερότητα. Να μην λέμε ελεύθερο εμπόριο, να λέμε καλύτερα θεμητό εμπόριο, δίκαιο εμπόριο, fair trade γιατί το ελεύθερο εμπόριο νοείται μεταξύ ισότιμων εταίρων. Αν μιλούμε για ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Ένωσης και αναπτυσσόμενων χωρών, είναι λογικό ότι ο ισχυρότερος εταίρος θα καρποθεί τα ωφέλη εις βάρος του αναπτυσσόμενου. Όχι λοιπόν free trade, αλλά fair trade, όχι ελεύθερο, αλλά θεμητό, δίκαιο εμπόριο. Γιατί το ελεύθερο εμπόριο προϋποθέτει ισοτιμία και ελευθερία, κάτι που δεν ισχύει. Ο κύριος Ρόζενμπεργκ αναφέρθηκε επίσης ε, στο σημαντικό θέμα του περιβάλλοντος ή στο θέμα της ανάπτυξης. Δεν βοηθάει ούτε την αναπτυξιακή μας, ούτε τη μεταναστευτική μας πολιτική. Αν εξάγουμε ταυτόχρονα οπλισμό προς αναπτυσσόμενες χώρες ή μειώνουμε τον πλούτο ορισμένων αναπτυσσόμενων χωρών εξαιτία της γεωργικής μας ή της αλληλευτικής μας πολιτικής. η στο θεμα της αναπτυξης δεν βοηθαει ουτε την αναπτυξιακη μας ουτε τη μεταναστευτικη μας πολιτικη αν εξαγουμε ταυτοχρονα οπλισμο προς αναπτυσσομενες χωρες η μειωνουμε τον πλουτο ορισμενων αναπτυσσομενων χωρων εξαιτια της γεωργικης μας η της ελλειφτικής μας πολιτικης αν ε, εφαρμόζουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, όπου ουσιαστικά στέλνουμε ναι, υλικά προς τη Σαχάρα για εκμετάλλευση, αλλά καρπονόμαστε εμείς οι ίδιοι την ενέργεια. Άρα τον πλούτο που δίνουμε τον παίρνουμε πίσω και δεν αφήνουμε τίποτα για την περιοχή. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τις επιπτώσεις των πολιτικών μας. Το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και εδώ θα πρέπει να ληφθεί περισσότερο υπόψη, γιατί σε πολλές χώρες βλέπουμε αυτή την τάση της προσέγγισης ε, των μεταναστών με βάση το πόσο επικερδής θα είναι για την ε, οικονομία, πόσο χρειάζονται για να καλύψουν κάποια κενά της αγοράς εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι οι μετανάστες είναι ανθρώπινα όντα, με ανθρώπινα δικαιώματα, όπως το να φύγουν από τη χώρα τους, να ζητήσουν άσυλο, να τύχουν προστασίες. Αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά όχι μόνο της μεταναστευτικής αλλά και της αναπτυξιακής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάουρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Προβέρα και την Κρέτου γιατί επέτρεψα να γίνει αυτή η συζήτηση για τη μετανάστευση. Θα ήθελα τη γνώμη των ομιλητών και πιο συγκεκριμένα από τον καθηγητή Μπρινέ. Ίσως λένε ορισμένοι το πρόβλημα της Ευρώπης σήμερα είναι η έλλειψη μιας πραγματικής ευρωμεσογειακής στρατηγικής. Όλες οι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από τη διαδικασία της Βαρκελόνης έχουν, <clears throat> θα έλεγα, δεν έχουν μάλλον τα απαιτούμενα μέσα τα οποία χρειάζονται και τα οποία μας έχουν κάνει την περιγραφή, για τα οποία μας έκαναν την περιγραφή οι ομιλητές. Υπάρχουν ε, βέβαια ορισμένοι αριθμοί με, ανησυχητικοί σχετικά με τις δημογραφικές αυξήσεις, όπως επίσης και τις οικονομικές βελτιώσεις των χωρών του Μαγκρέμπ. Από την πρώτη ανάγνωση διαπιστώνει κανείς ότι οι δύο δρόμοι που έχουμε στη διάθεσή μας, από τη μία δηλαδή να ευνοήσουμε την οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση των οικονομιών αυτών των χωρών και από την άλλη να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές, φαίνεται ότι και οι δύο αυτοί δρόμοι από μόνοι τους δεν λύνουν το πρόβλημα. Έχει δίκιο ο καθηγητής Μπρινέ όταν λέει ότι τη στιγμή που αυξάνεται, που βελτιώνεται η οικονομία των χωρών αυτών, υπάρχει η δημογραφική ανάπτυξη των χωρών αυτών, που καθιστά θα έλεγα περιτά ε, τα αποτελέσματα τα θετικά της οικονομικής ανάπτυξης στη μετανάστευση. Ακόμα και αν αυξήσουμε λοιπόν ε, τους πόρους για την ανάπτυξη στις χώρες αυτές, δεν λύνουμε τα προβλήματα χωρών όπως η Τινησία, η Αλγερία και το Μαρόκο. Γι' αυτό θα ήθελα να μου πει ο κύριος Μπρινέ ποιο είναι το σωστό μίξ που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε σε μια ελεγχόμενη μετανάστευση αυτών των χωρών και ποια θα είναι τα ποσοστά τα οποία θα πρέπει να επιλέξουμε για τις πολιτικές αυτές τις ανάμεικτες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν βέβαια τις οικονομίες των χωρών. Ακόμα και αν επενδύσουμε λοιπόν στην οικονομική ανάπτυξη χωρών σαν το Μαρόκο, μπορεί να έχουμε σαν συνέπεια ένα φαινόμενο ισχυρού ανισμού με τις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία σαν παράδειγμα, κάτι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχικυκλώματα θα έλεγα στην ευρωμεσογειακή πορεία. Λοιπόν, περιμένω από τον καθηγητή Μπρινέ να πει ποιο είναι το σωστό μίξ σε εισαγωγικά. Ε, πώς μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε ε, και σε ποιο βαθμό τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Δύσκολη ερώτηση. Πρώτα θα μιλήσει ο κύριος Μπεναβέντε, μετά ο κύριος Μπρινέ και φυσικά όποιος από τους ομιλητές εδώ θέλει να πάρει το λόγο τον έχει. Ευχαριστώ. Άκουσα μια ερώτηση, αλλά δεν είμαι αρμόδιος για να απαντήσω. Με ρωτήσατε γιατί κάποιες χώρες μέλη δεν ε, κυρώνουν την συνθήκη για την προστασία των μεταναστών και των οικογενειών τους. Φαντάζομαι ότι αυτό οφείλεται σε θέματα εσωτερική του νομοθεσία. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω την παρέμβαση της κυρίας Κέλλερ. Δηλαδή, να μην χορηγήσουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε χώρες διέλευσης. Συμφωνώ απόλυτα. Οι χώρες διέλευσης είναι και η σχέση με αυτές καλύτερα να αντιμετωπιστούν θέματα διμερών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής. Free trade και fair trade. Συμφωνώ και με αυτό το σχόλιο. Um, merci, uh, monsieur. Ο κύριος Μπρινέ. Σύμφωνο, ε, σας ευχαριστώ θερμά για τις ερωτήσεις σας. Σε ό,τι φορά τη χορήγηση ή όχι αναπτυξιακής βοήθειας στις χώρες διέλευσης, αν ε, λάβουμε το παράδειγμα της Λιβύης, γιατί είναι όντως χώρα διαέλευσης και όχι χώρα προέλευσης της μετανάστευσης, πέραν της συνεργασίας που έχουμε για τον έλεγχο στα σύνορα, για τον οποίο έλαβα υπόψη και αντιλαμβάνομαι τις παρατηρήσεις δεδομένου ότι δεν έχουμε εθνικό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των μεταναστών, και δεδομένων των συνθήκων κράτησης των ελαφρομεταναστών ή και λήψη πολιτικής οργάνωσης της νόμιμης μετανάστευσης στη Λιβύη, είναι ανάγκη, πιστεύω, η Ευρωπαϊκή η Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψουν μια εταιρική σχέση και να έχουν ένα πολιτικό διάλογο με τη χώρα αυτή, παρέχοντας τεχνογνωσία ή τεχνική αρρωγή, προκειμένου και η Λιβύη να εφαρμόσει ένα σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων ή των ετούντων άσυλο και να βελτιωθούν οι βιωτικές συνθήκες των μεταναστών. Είναι θέματα ανθρωπιστικού δικαίου και νομίζω ότι είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιμείνει σε αυτή την κατάσταση, να εμπλακεί, γιατί δεν μπορούμε να θελοτυφλούμε απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα αυτή και στη μεταχείριση των μεταναστών εκεί. Δεν λέμε να δώσουμε μόνο χρήματα στη Λιβύη για να ελέγξει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα ήταν μια πολύ κοντόφθελμη ε, προσέγγιση σε ό,τι αφορά το αίτημα του Συμβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία με τη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κυρίου Μάουρο για την σωστή ισορροπία πολύ δύσκολη ερώτηση, μάλλον ρητορική. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ταυτόχρονα και τους δύο πυλώνες. Δηλαδή, για λόγους συνέπειας με τους στόχους της αναπτυξιακής μας πολιτικής, αλλά και για οικονομικούς λόγους, θα πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη των χωρών Μαγκρέπ. Εκτός του ότι οι χώρες αυτές είναι και σημαντικές αγορές για τις επιχειρήσεις μας, υπάρχουν και προφανείς λόγοι που συνηγορούν υπέρ της ανάπτυξης ε, της γεωργίας ή των θέσεων εργασίας στη γεωργία και υπάρχουν ε, πολλές ευκαιρίες ε, για αμοιβαία επωφελή σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο εταίρων. Έχουμε ανταγωνισμό στην κλωστή φαντουργία με την Κίνα και την Ασία γενικώ και από αυτήν την άποψη πιστεύω ότι με τις χώρες του Μαγκρέφ θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε εταιρικέ σχέσεις στην κλωστή φαντουργία. Και αυτό κάνουν τόσοι ή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, οι ιταλικές, οι ισπανικές. Και δεν είναι τυχαίο που μετεγκατέστησαν τα εργοστάσια τους στο Μαγκρέμπ. Εκεί βρήκαν ευκαιρία για ανάπτυξη αμοιβές, επαναλαμβάνω υποφελών εταιρικών σχέσεων και για τις χώρες της περιοχής και για το Μαγκρέπ και για τις ε, επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο να αναπτύξουμε την νόμιμη μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Ναι, αυτό κάνουν ε, και πολλές χώρες με Δείτε τις συμφωνίες εργατικού δυναμικού μεταξύ Ιταλίας και Τινησίας, ή Ισπανίας και Μαρόκου και πρόσφατα μεταξύ Γαλλίας και Τινησίας διαπιστώνουμε ότι εκεί υπάρχει ένα αναπτυξιακό δυναμικό μίας νόμιμης μετανάστευσης που θα καλύψει τις ανάγκες αγοράς εργασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα, πλαισιώνοντας και κατοχυρώνοντας τα δικαιώματα των μεταναστών που καλύπτονται από αυτές τις συμφωνίες εργατικού δυναμικού. Νομίζω ότι όλες αυτές τις πτυχές θα μπορούσαμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω, γιατί υπάρχουν ανάγκες στην αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαίνεται και από τις δημογραφικές προβλέψεις. Μέχρι το 2050 θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τεράστιες ανάγκες ειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Γι' αυτό και οι χώρες Μαγκρέπ από την άποψη είναι η φυσική μας εταίρη για την ανάπτυξη μιας νόμιμης μετανάστευσης. Ha chiesto di intervenire il signor Ζήτησε το λόγο ο κύριος Ρόζενμπουργκ. Um, thank you. Um, yeah, two remarks. One on, on migrant rights. Um, as you know, earlier this Δύο παρατηρήσεις. <clears throat> Αυτή την εβδομάδα οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων Αφρικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν στην Τρίπολη και συμφώνησαν σε μια νέα εταιρική σχέση μια νέα εταιρική σχέση που έχει και ένα σκέλος στον τομέα της μετανάστευσης. Το θέμα δεν είναι αυτό βέβαια, το θέμα είναι ότι στα πλαίσια αυτή της εταιρική σχέσης ένα βασικό κομμάτι της πολιτικής είναι η επιβεβαίωση θα έλεγα τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τα δικαιώματα των μεταναστών, τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Στα πλαίσια αυτή της πολιτικής θα υπάρξει διάλογος και συνεργασία και αυτό είναι πρώτη φορά που γίνεται. Αυτό αφορά τους μετανάστες στην Ευρώπη αλλά φυσικά και στην Αφρική. Γιατί εκεί είναι η μεγαλύτερη ομάδα θα έλεγα και έτσι θα μπορέσουμε πλέον να συζητήσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών στη Λιβύη ή σε άλλες χώρες της Αφρικής που μπορεί να απειλούνται. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σημαντικό πολιτικό βήμα και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε ε, να περάσουμε σε θετικά αποτελέσματα για την ε, ερώτηση Λόχμπιλερ για το μέγεθος των μεταναστευτικών ροών που προκαλείται από τις κλιματολογικές αλλαγές και τη χειροτέρευση του κλίματος γενικότερα. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να συλλέγει αριθμούς τέτοιου είδους. Εμείς επαφιέμεθα στη στοιχεία που δίνουν είτε διεθνείς οργανισμοί είτε εθνικοί οργανισμοί και δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω λοιπόν το συγκεκριμένο. Πάντως, ακόμα και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την δυνατότητα γενικότερα και ξεκινάμε σε ένα μήνα ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ στα πλαίσια του Ταμείου Ανάπτυξης ε, για το παρατηρητήριο των μεταναστεύσεων το οποίο θα μας επιτρέψει στο μέλλον να έχουμε καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στη συνάδελφο Κρέτου για να κλείσει τη συζήτηση, Α, για, συγγνώμη, η κυρία Πάτσε έχει ζητήσει το λόγο, ζητώ συγγνώμη, δεν ήθελα να σας αποκλείσω. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω κάποιες από τις ερωτήσεις που τέθηκαν σχετικά με τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στη μετανάστευση. Λυπάμαι που δεν έχω, θα έλεγα, πολλά αντίτυπα από το βιβλίο αυτό το οποίο περιλαμβάνει ε, στοιχεία. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, εκτιμήσεις από λίγα εκατομμύρια σήμερα να περάσουμε σε πολύ περισσότερα εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Πάντως ε, είναι σαφές ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του φαινομένου και επί τη βάση των στοιχείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ήθελα εδώ ότι έχουμε κάνει μία μελέτη για το Κοινοβούλιο ε, για τη μετανάστευση στις 27 χώρες, κάτι που είναι διαθέσιμη Έχουμε κάνει επίσης ε, και μία μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών σχετικά με τις επιπτώσεις της μετανάστευσης. Αυτά θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σχετικά με την ερώτηση που τέθηκε για την προστασία των μεταναστών, υπάρχουν κάποιες, κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε εδώ στη διάθεσή μας, όχι νομικού τύπου αλλά πολιτικού τύπου. Είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να γίνουν αντικείμενο περαιτέρω δουλειάς και υπήρξε και μία μελέτη της UNESCO που έκαναν δύο παλαιότεροι συνάδελφοί μου Λοιπόν, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον άλλο, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τη γνώμη σας τώρα σχετικά με μια κατάσταση η οποία συναντάται θα έλεγα σε όλες τις υπήρους. Δηλαδή την εσωτερική μετανάστευση σε μια ήπειρο, σαν παράδειγμα στην Αφρική. Έχουν υπάρξει αφρικανικές χώρες οι οποίες είναι αντικείμενο θα έλεγα μεταναστευτικών ροών όπως η Λιβύη και στα πλαίσια της πολιτικής που ξεκίνησε εδώ και λίγα χρόνια του Παναφρικανισμού δηλαδή από τον Καντάφη. Έλεγε ουσιαστικά ότι ο κάθε Αφρικανός είναι και πολίτης της Λιβύης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους Αφρικανούς πολίτες λοιπόν να μεταναστεύσουν να θέλουν και να γίνουν κάτοικοι της Λιβύης. Αυτό δημιούργησε ένα σοβαρό πρόβλημα στη Λιβύη το οποίο ε, εν μέρη εκτονώνεται με τη μετανάστευση προς την Ευρώπη. Λοιπόν, στον τομέα αυτό λέει ο, ο μιλητής, όλα είναι αλληλοεξαρτημένα. Υπάρχουν μελέτες ε, και σε σχέση με τις δυνατότητες οικονομικής βοήθειας ε, σε περιφερειακό επίπεδο στις χώρες αυτές και αν ναι με ποια μέσα. Μια δεύτερη ερώτηση πιο απλή. Χρησιμότητα μιας μόνιμης δομής ε, διαιτησίας των συγκρούσεων τουλάχιστον για τις γειτονικές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να αποφύγουμε μελλοντικές περιοχές νέας κρίσης. Ευχαριστώ. ο κύριος Μπρινέ για την πρώτη σας ερώτηση. Θα ήταν χρήσιμο να αναπτύξει κανείς τους μηχανισμούς και τα μέσα για την τριγωνική λεγόμενη συνεργασία ανάμεσα σε ορισμένες από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και τις χώρες της υποσαχαρικής Αφρικής. Έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις αλλά πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Και υπάρχει η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο δραστήρια στα πλαίσια αυτής της τριγωνικής ε, συνεργασίας. Οι χώρες αυτές αναπτύσσονται βέβαια και ενδιαφέρονται και για την ανάπτυξη των γειτονικών τους χωρών. Ας πούμε οι χώρες αυτές ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των χωρών Σαέλα, της υποσαχαρικής δηλαδή ε, περιοχής αναγνωρίζουν την ανάγκη επένδυσης όχι μόνο στην ασφάλεια των συνόρων τους, αλλά και στην ανάπτυξη γενικότερα των γειτονικών χωρών. Υπάρχει λοιπόν μια δυνατότητα εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζεται άμεσα Όσο εκ τούτου λοιπόν έχουμε κοινά συμφέροντα χώρες του Μαγκρέμπ και ευρωπαϊκές χώρες να αναπτύξουμε περισσότερες δράσεις και για να το πετύχουμε απαιτείται να έχουμε στη διάθεσή μας τα μέσα για να επηρεάσουμε την κατάσταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Βόρεια Αφρική και στην υποσαχαρική Αφρική. Προ στιγμή τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι τα καταλληλότερα Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης της παρέμβασής μας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρόζενμπουργκ. Έχει σημασία να δούμε και τι κάνει ο Οργανισμός Αφρικανικής Ενότητας. στα πλαίσια και της περιφερειακής μορφής αυτής συνεργασίας και στα πλαίσια των οικονομικών κοινοτήτων της Αφρικής. Όλοι προσπαθούν να προωθήσουν την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στις χώρες τους. Όλες οι χώρες αυτές έχουν ε, πρωτόκολλα διμερεί και τα οράματά τους όταν συζητάμε μαζί τους είναι να χρησιμοποιήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν παράδειγμα σε σχέση με την ελεύθερη διακίνηση. Βέβαια, αν τυχόν μπορεί κανείς να βρει μια θέση δουλειά στη χώρα του με εύκολο τρόπο και με καλές συνθήκες, σεβασμού δικαιωμάτων κτλ, ε, τότε δεν υπάρχει λόγος να σκεφτεί κανείς τις εναλλακτικές λύσεις όπως ε, η μετανάστευση. Και η κυρία Κρετού για να κλείσει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις σας. Ήταν ε, μεγάλη τιμή για μας να ενημερωθούμε τόσο σωστά για αυτό το σημαντικό θέμα που αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια γύρω από αυτά τα, τις, τα, τις τρεις διόδους βέβαια. Σχετικά με τη λεγόμενη φυγή των εγκεφάλων θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και την έλλειψη ανθρωπίνων πόρων ιδιαίτερα στις χώρες προέλευσης το αποτέλεσμα των εμβασμάτων, θα έλεγα του φαινομένου των εμβασμάτων που επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης, χρησιμοποιείται φυσικά το φαινόμενο αυτό σαν μέσο βοήθειας οικονομικής. Ο κύριος Μάουρο δεν είναι ακόμη εδώ. Αλλά είναι προβλήματα όλα αυτά και φαινόμενα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Και είναι και ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο γιατί από τις χώρες ε, προέλευσης, ε, σαν παράδειγμα, στις χώρες προέλευσης ε, εισέρχονται πάρα πολλά εμβάσματα από τους μετανάστες που έχουν πάει στις χώρες που τις φουλεξενούν σήμερα. Σε επίπεδο αναπτυξιακό νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τα χρηματοδοτικά αναπτυξιακά μέσα το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο και την ανθρωπιστική βοήθεια βέβαια, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τους λεγόμενους πρόσφυγες ε, της πείνας. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, αν και έχουμε αρκετά προγράμματα στη διάθεσή μας. Και τέλος, νομίζω ότι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία στις πιο εύθραστες, ευάλωτες ομάδες μεταναστών, τις γυναίκες και τα παιδιά. Η αρχή της έλλειψης διακρίσεων πρέπει να εφαρμόζεται και στην πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας και θα πρέπει τα θεμελιώδη δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά. Τα παιδιά τα οποία μεταναστεύουν θα πρέπει να γίνονται και αυτών τα δικαιώματα σεβαστά. Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Ελπίζω να έχουμε την δυνατότητα η συζήτηση αυτή να ξαναγίνει και σε εμά και στην Ολομέλεια για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ευχαριστώ κυρία Κρέτου. Περνάμε στο δεύτερο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον Πέτερ Φάιντα τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσφοπέδιο. Αλλά χρειαζόμαστε λίγα λεπτά. Grazie molto, thank you very much. Thank you, merci monsieur. Ciao.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 Bene. Proseguiamo con il punto seguente. Συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο. Και όμως σας είπα ήδη, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βίτερ Φάιτ, αδικό αντιοτελμένο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κουσιβοπαίδιο. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας καλωσορίσω, κύριε Φάιτ, που είναι συχνός επισκέψεις της Επιτροπής αυτής και σήμερα θα μας παρουσιάσετε τη μαρτυρία της σε μια πολύ λεπτή φάση της ε, ζωής στο ψυχοπαίδιο ενώπιση των εκλογών της 12 η Δεκεμβρίου. και της ε, μονομερούς ε, δήλωσης της χώρας αυτής. Ε, θα υποστείλουμε μία αποστολή παρακολούθησης των εκλογών και αυτό είναι σωστό να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική διαδικασία. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον κύριο Φάιτ για την υποστήριξη που δίνει στην ε, αποστολή αυτή. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω μέσα στο λόγο για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. To uh, be again um, in this committee under your leadership. Είναι μεγάλη μου τιμή που μπορώ να είμαι εδώ. To the European. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή του Κοινοβουλίου στην εξέλιξη στην ε, στο Πεσικοπαίδιο, ως ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου, θα έλεγα ότι πραγματικά γίνεται αισθητή η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφέρων που αποδίδουν επιτόπου. Και αυτό ενδυναμώνει σημαντικότατα την ευρωπαϊκή φωνή στο Πέδιο. Ο ασκόντο καθήκοντα του Προέδρου κ. Κόσνουστη κάλεσε επίσημα μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρακολουθήσει τις επερχόμενε εκλογέ. Και χαίρομαι που 7 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έρθουν σε μια επίσημη ε, αντιπροσωπεία στην ημέρα των εκλογών, στις 12 Δεκεμβρίου. Ένα σημαντικό Μέσω υποστήριξης θα είναι αυτό και το πόρισμα της αντιπροσωπείας θα ε, βαρύνει πάρα πολύ την άποψη και στην περιοχή και εκτός. Ταυτόχρονα η επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα της ε, η για το κοσμοπέδιο της κυρίας Λούνασεκ ήταν καλό δεκτή και ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Στην ε, κοινή μας επίσκεψη μπορέσαμε να μεταβιβάσουμε μηνύματα αλλά και να κάνουμε και επικρίσεις και να δώσουμε την πιο ευρεία ευρωπαϊκή προοπτική αναφέροντας βέβαια την ανάγκη να γίνει σεβαστή η πολιτιστική κληρονομιά που είναι τόσο σημαντική για τις ευρωπαϊκές αξίες που προσπαθούμε να υποστηρίξουμε. Η επίσκεψη έδειξε μεγάλη ενδιαφέροντος και προσοχής στα ΜΜΕ. Η κυρία Λούνατσεκ επισκέφθηκε επίσης το βόρειο κοσυβοπαίδιο ε, καταδεικνύοντας την υποστήριξη του Κοινοβουλίου όλων των κοινοτήτων του κοσυβοπαιδίου. Πρόσφατα κύριε Πρόεδρε είδαμε μία σειρά σημαντικών προφανώς εξελίξεων στο κοσυβοπαίδιο και γύρω από το Καταρχήν, ε, οι επερχόμενες εκλογές, η έκθεση πρόεδρος της που προετοιμάζεται, ε, η υποστήριξη της ε, απελευθέρωσης των θεωρήσεων των διαβατήριων και οι συνεχόμενες μας προσπάθειες να αποδώσουμε σημασία στις επερχόμενες συζητήσεις με τη Σερβία. Όλα αυτά τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ σημαντικά και αποδεικτικά στοιχεία του αυξανόμενου ρόλου του, της Ευρώπης στο κωσυφοπαίδιο. Θα μου επιτρέπετε να αναφερθώ στις εκλογές που βέβαια κυριαρχούν τις πολιτικές αυτή τη στιγμή στο κωσυφοπαίδιο. Μετά την διάλυση της Βουλής του Κωσυφοπαίδιου ορίστηκαν πρόορες εκλογές στις 12 Δεκεμβρίου. Αυτές είναι οι πρώτες γενικές ε, εκλογές που οργανώνονται από τα νέα θεσμικά όργανα του Κωσυφοπηδίου. Είναι μια σημαντική ευκαιρία να καταδειχθεί η ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Παρόλο το σύντομο του χρόνου έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τις εκλογές. Μία εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών έχει ξεκινήσει και θα μπορεί παραντονιστεί η σημασία συμμετοχής όλων των κοινοτήτων. Η υπηρεσία μου έχει υποστηρίξει πολλές ε, οργανώσεις των πολιτών για να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των μειονοτήτων, ε, των νέων και όλων των ομάδων Οι Η και οι ε, προετοιμάζονται να κρατήσουν την τάξη μαζί με την ε, αστυνομία του Κωσυφοπεδίου. Ιώσε, δεν θα παρατηρήσει ακριβώς τις εκλογές την ημέρα των εκλογών, αλλά εργάζεται στην προετοιμασία. Η υπηρεσία μου θα συντονίσει αυτό που αποκαλούμε διπλωματική, διπλωματικό παρατηρητήριο των εκλογών, Εκατό ομάδες επισήμων, υπαλλήλων, διπλωματών από τους δικούς μας ε, υπηλήλους ε, από τις πρεσβείες και άλλες οργανώσεις και Πριστινά και αλλού στην περιοχή. Και θα ήθελα εδώ να σημειώσω την ευγνωμοσύνη μου προς τα κράτη-μέλη για την ε, σαφή τους υποστήριξη. Ήταν πάρα πολύ θετικά όσον αφορά τον ρόλο της USR και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα προς το ξεφοπέδο τις ε, σημασία που αποδίδεται στην κατάσταση δημοκρατισμού του Κωσυφοπαθείου. Προσβλέπουμε βέβαια να έχουμε την επίσημη σας ε, ε, αντιπροσωπεία εκεί. Υποθέτω ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι στον συνασπισμό δύο κοσοβοαλβανικών κομμάτων. Αν γίνει αυτό, αυτό θα σημαίνει ισχυρή βάση για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις που επίκειται. Στα μήνυματά μου προς τα ηγέτες των κομμάτων είπα ξεκάθαρα ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια καθαρή κυβέρνηση. Ειλικρινά, όπως το ξέρουμε, έχουν πρόγραμμα, πρόγραμμα εικόνας που παρουσιάζουν και το κοσμοπέδιο και οι ηγέτες τους και αυτό θα πρέπει να σταματήσει η κυβέρνηση θα πρέπει να είναι όχι μόνο καθαρή, αλλά και ικανή. Γιατί υπάρχουν ουσιαστικότατες προκλήσεις, μία εκ των οποίων είναι οι κοινωνικο-οικονομικές προϋποθέσεις της χώρας. Βλέπουμε βραδία ανάπτυξη που βασίζεται κυρίως σε δημόσιες επενδύσεις. Η ανεργία είναι στο διπλάσιο του μέσου όρου της περιοχής. Ο μέσος όρος εισοδημάτων χαμηλός και υψηλά ποσοστά ένδυας. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να βελτιώσει το περιβάλλον για επιχειρήσεις και για επενδύσεις. Αυτό σημαίνει δομικές αλλαγές στην ενέργεια, ορυχεία και τηλεπικοινωνίες. Σημαίνει μία ε, ε, σταθερή και ε, συνετή πολιτική στον τομέα το φορολογικό και η κράτος δικαίου. Αυτή η καθαρή και ικανή νέα κυβέρνηση με νέες ιδέες θα είναι καλή προϋπόθεση, προϋπόθεση για να συνεχιστεί πρόοδος στις σχέσεις του Κωσυφοποδίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το κύριο θέμα θα είναι εδώ είναι ε, διευκολυμένος ε, διάλογος μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Σερβία. Εκλογές σημαίνουν βέβαια ότι αυτός ο διάλογος δεν μπορεί παρά να αρχίσει μετά τις εκλογές, κατά πάση μετά μάλιστα μετά την ενέξη του νέου τους. Όμως φαίνεται ότι είναι έτοιμο να δεσμευθεί το κοσυβοπαίδιο και καλύτερη συνεννόηση μεταξύ Βρυξελών και Ουάσιγκτον έδωσε πολύ εμπιστοσύνη στους Κωσοβάρους και στους ηγέτες τους. Υπάρχουν πολλές ανησυχίες βέβαια για την διαδικασία αυτή. Οι Κωσοβάροι ε, δέχονται ότι υπάρχουν αυτές οι κόκκινες γραμμές, αλλά υπάρχουν και οι γαλάζιες γραμμές θεμάτων που ανησυχούν όλους τους πολίτες. Θέματα που δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη λειτουργία του κράτους σε τομείς όπου υπάρχει αυτή τη στιγμή μπλοκάρισμα θεμάτων. Και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, πρόοδο σε, σε τομείς όπου η Σερβία θα έπρεπε λόγω των ε, δεσμών που έχει με το κοσυφοπέδιο, συγγνώμη, οι δεσμοί αυτοί όμως έχουν κάπως καλυφθεί. Είμαι πεπισμένος κύριε Πρόεδρε ότι είναι δυνατή η πρόοδος. Το καθοριστικό θέμα για τη χώρα και για την ε, διεθνή κοινότητα είναι το βόρειο κοσυφοπαίδιο. Υπάρχουν σημαντικότητε προκλήσεις εδώ. Θα ήθελα όμως να επιστήσω την προσοχή σας στην τη πρόοδο που παίζει Ε, ο, παίζει το, το, κέντρο του κοσμοπέδιου στο υπόλοιπο της χώρας. Είχε ελεγχθεί στο παρελθόν ότι δεν επρόκειτο να ενδεσμευθούν και να συμμετάσχουν στις τοπικές αυτοδικήσεις της περιοχής εκείνης οι Σέρβοι. Όμως το αντίθετο συνέβη. Βέβαια δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί η εργασία, αλλά είναι θετικό σημείο ότι βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση το κοσυφοπέδιο. Και σκέφτομαι εδώ ε, όπως όπως Σκρατσανίτσα και Σρέψε. Και οι δήμαρχοι τους είναι απόλυτα δεσμευμένοι να λειτουργήσει σωστά το Κόσοβο για αυτούς. Ο καθένα θα πρέπει να ψηφίσει για να δει τι θα γίνει τελικά. Ακριβώς τη Δευτέρα συνάντησα τους ηγέτους μιας νέας σερβικής πολιτικής ομάδας που θα συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές. Αυτοί περιμένουν αυξημένη σερβική συμμετοχή. Το βόρειο κοσυβοπαίδιο αλλάζει επίσης. Και την ίδια αλλαγή που είδαμε να λαμβάνει η χώρα στο νότο θα είναι δυνατόν να τη δούμε και στο βορρά. Βέβαια τα πράγματα δεν θα αλλάξουν γλίγορα, ούτε εύκολα. Υπάρχουν Σέρβοι στο βορρά που θέλουν να συμμετάσχουν πολιτικά, αλλά είναι θύματα βίας από εκείνους που θέλουν να παραμείνει στάσιμη η πολιτική κατάσταση. Υπάρχουν επίσης ε, Κωσοβοσέρβοι στο βορρά που θέλουν να δεσμευτούν οικονομικά. Αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους εγκληματίες και να ε, προωθήσουν το κράτος δικαίου. Αυτό απαιτεί τόλμη, θάρρος, αλλά και μια κυβέρνηση Κωσοπεδίου που είναι πρόθυμη να προστατεύσει μια μειονότητα με λόγια και με πράξεις. Χρειάζονται δημοκρατικές επιλογές και οικονομικές ευκαιρίες οι κάτοικοι του Κωσοφοπεδίου δεν τις έχουν αυτή τη στιγμή και δεν θα είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι όλοι ξαφνικά θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις εκλογές. Αλλά από την άλλη μεριά δεν θα πρέπει να υπάρχει ανοχή για ε, πράξεις εκφοβισμού. Επιτροπή σας ε, χθες ζήτησε ακριβώς την καταστροφή των παραλλήλων δομών στο Κωσυφοπαίδιο και αυτό το χαιρετίζω ιδιαίτερα. Πολιτιστικά και θρησκευτικά θέματα εξακολουθούν να είναι κεντρικά της προσοχής μου. Και χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι και εδώ υπάρχουν μηνύματα ε, πρόοδου. Ο Έλληνας πρέσβης Δημήτρης Μοσχόπουλος ε, δρά έντονα στην, στον τομέα αυτόν. Ο νέος πατριάρχης ε, της ε, Σερβικής Ορθοδοξής Εκκλησίας με ασφάλεια και ο ανθρωπισμός του με ασφάλεια που προσέφερε η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου σε συντονισμό με την EULEX απέστειλε επίσης ένα σημαντικό θετικό μήνυμα. η μεταφορά από την προστασία του ΚΑΦΟ στην αστυνομία του Κωσυφοπεδίου ορισμένων αυτών των θρησκευτικών ε, ε, τοποθεσιών προχωράει πολύ καλά. Σε Σόβρο που είχα πάει με την κυρία Νόντσεκ ακούσαμε θετικά θέματα όσον αφορά την επιστροφή Σέρβων και την αναζωογόνηση της ε, θρησκευτικής κοινότητας και ενδεχόμενη μάλιστα προσαγωγή ε, μοναχών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει. Η ρόλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προσδοκίες θα πρέπει να επιδράσουν και στο Βελιγράδι και στην Πριστίνα. Βασικές ευρωπαϊκές ιδέες δημοκρατίας, ασφάλειας και οικονομικών ευκαιριών δεν είναι λειτουργικές σε, αυτό το, σε αυτή τη μικρή περιοχή του Κωσυφοπεδίου. Και η Ulex είναι εκείνη που αρχίζει να μεταστρέφει τα πράγματα. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης στις προσπάθειες πιο ευρείας διεθνούς ε, κοινότητας να έχει πρόσβαση εκεί για σχέδια προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης των πολιτών του Βορείου Κωσυφοπεδίου. Επίσης θα ήθελα να τονίσω μετά από συζητήσεις με τόπιους ότι ακόμα και εκείνοι που παραμένουν αβέβαιοι όσον αφορά το θέμα της ανεξαρτησίας του Κωσυφοβιδίου είναι 100% σίγουροι ότι θέλουν βασική ασφάλεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ο διευκολυμένος διάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να προωθήσει τη διαδικασία ε, ομαλοποίησης. Κύριε Πρόεδρε, σοφά ελέγχθη ότι η διαδικασία του διαλόγου αφορά την προσέγγιση και τη εργασίας του Κωσοβοδίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θε, πρέπει να δούμε και οι μεν και οι δε να κάνουν συγκρίσιμα βήματα ακόμα και αν βρισκούν σε διαφορετικά στάδια του ταξιδιού. Αλλά όλα αυτά ούτε δωρεάν είναι ούτε εύκολα. Η πρόσφατη έκθεση προόδου της Κομισιόν για το Κωσυφοπαίδιο ήταν μια ισορροπημένη και καλή παρουσίαση. Υπάρχει σημαντική πρόοδος στην αποκέντρωση, στο σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και στις, στην αστυνομία. Υπάρχουν όμως σημαντικοί τομείς όπου χρειάζεται πραγματικά περαιτέρω εργασία, συμπεριλαμβανομένως της καταπολέμησης της διαφθοράς, ενδυνάμωσης του τμήματος δικαιοσύνης, του δικαστικού, και πλήρη σεβασμός της ελευθερίας του τύπου. Η Πρίστινα περνάει μια σημαντική διαδικασία εκμάθησης με το θέμα της απελευθέρωσης της θεώρησης ε, διαβατηρίων. Ο διάλογος για το θέμα αυτό δεν είναι κάτι που είναι βραβείο για καλή συμπεριφορά. Υπάρχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες τεχνικές απαιτήσει. Το παιδί, τώρα αρχίζει να το κατανοεί. Κατανοεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια κοινότητα κρατών μελών με πάρα πολλές πραγματικές και πρακτικές ανησυχίες. Στο θέμα αυτό, σας λέω πραγματικά ότι στην αρχή υπήρχε μία έκπληξη και απογοήτευση από την Πριστίνα. Πιστεύουν επίσης ότι η διεθνής κοινότητα θα έπρεπε να έχει μετατεθεί περισσότερο μετά από την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηριού ότι η δήλωση ανεξαρτησίας δεν ήταν ε, ενάντια στον διεθνή νόμο. Στο Κωσυμπεπέδιο πιστεύουν ότι τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα στην πλήρη αναγνώριση ε, της ανεξαρτησίας τους δεν πρέπει να παραβλέπετε. Πιστεύουν ότι χρησιμοποιούν δύο μέτρα και δύο σταθμά για αυτούς και τους γειτονές τους. Πρόσφατα, σε βολιδοσκοπήσεις που έγιναν, ο αριθμός των ε, Κωσοβάρων που πιστεύουν ότι δεν τη χάνουν σωστή συμπεριφορά έπεσε στο 10%. Ξέρουμε το κίνδυνο του να αφήσουμε στον εθνικισμό και στον σκεπτικισμό μεγάλα περιθώρια δεν μπορούμε να επιτρέψουμε το αίσθημα της ε, αποτελμάτωσης και της απομόνωσης να συνεχιστεί, να εδραιωθεί. Είδαμε όμως και αλλού στα Βαλκάνια ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφής, η, η δημόσια κατανόηση είναι σαφής και η στόχη είναι σαφής, τότε μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Εάν πιστεύουμε ότι έχουμε συμφέρον ως κράτη-μέλη και ένωση να δούμε σταθερότητα και πρόοδο στο ψηφοπαίδιο, τότε πιστεύω ότι έχουμε συμφέρον να παραμείνουμε θετικοί και ρεαλιστές. Ελπίζω ότι χωρίς να προδώσουμε τις βασικές μας αρχές, θα εξακολουθήσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες ώστε το Κωσυφοπαίδιο να, πε... να πλησιάσει περισσότερο ένα ευρωπαϊκό περιφερειακό πλαίσιο. Το εμπόριο είναι ένα τομέα όπου η ανάπτυξη είναι καλή για όλου. Για το κοσυφοπαίδιο, για την περιοχή, για την ε, βούλησή μα να περάσουμε από τη βοήθεια σε πραγματικέ επενδύσει. Και ελπίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερο για να πάψουμε να μπλοκάρουμε την ε, δυνατότητα ε, εμπορίου του κοσυφοπαιδίου. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια θα πρέπει να παραμείνουμε συνεπείς και συνεκτική στα μηνύματα που θέλουμε. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς όσον αφορά τις επικρίσεις για μια χώρα όπως το Κωσυφοπέδιο. Θα πρέπει όμως να είμαστε σαφείς και όσον αφορά τις υποσχέσεις μας. Γιατί τα δύο εκατομμύρια πολίτες του Κωσυφοπεδίου αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή και λαμβάνουν πάρα πολύ σοβαρά και τις υποσχέσεις και τις επικρίσεις μας. Πρόεδρε, το Κωσυφοπέδιο δεν είναι πια θέμα ασφάλειας, είναι θέμα ανάπτυξης διακυβέρνησης, οικονομίας και κοινωνίας. Μετά τις εκλογές θα αναζητήσει οικονομική πρόοδο και ευρωπαϊκή πρόοδο. Θα πρότεινα να είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε αυτές τις δυνατότητες. Είναι προς όφελος και του Κωσυφοπεδίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο μεγαλύτερος ε, εταίρος του Κωσυφοπεδίου. Παραμένω πεπισμένο ότι το κοσυφοπαίδιο μπορεί και θα είναι επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ. Ήταν μεγάλη μου τιμή, το επαναλαμβάνω, και θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή που εξακολουθείτε να αποδίδετε στο κοσυφοπαίδιο και στα θέματα του κοσυφοπαιδίου. Προς τα παρόν προσβλέπω στις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ. Thank you Bene, eh, Καλώς. Έχουμε ένα μεγάλο κατάλογο ερωτήσεων. Η κυρία Λούνατσεκ, πρώτη εισηγήτρια. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Φέιθ για την ομιλία του. Συμφωνώ με ό,τι είπατε σχετικά με τον ρόλο κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την περιγραφή της κατάστασης στο Κοσμοπέδιο σήμερα. Αναφερθήκατε και στην επίσκεψη στο Πρίσβεν, έμαθα πολλά εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί ότι ανακαινίζεται ε, το τέμενος, το ίδιο θα γίνει και με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Ορθόδοξος Παπάς όταν πηγαίνει εκεί του λένε και καλημέρα. και γενικά υπάρχει μια κάποια ελπίδα για την αναγέννηση του Πρίζρεν, όπου κάποτε μιλούσαν και τρεις γλώσσες εκεί, γιατί υπάρχει και μια τουρκική κοινότητα στο Πρίζρεν. Υπάρχει κάποια ελπίδα. Ένα άλλο θέμα επίσης, το οποίο ήταν η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και είδα κάποιον που οργανώνει ένα φεστιβάλ ντοκιμαντέρς και υπάρχει ένα κινηματογράφος παλαιός από την εποχή της Ιουκοσλαβίας και θέλουν να τον χρησιμοποιήσουν και συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο. Και καλό θα είναι για την ιστορία του Πρίσβεν να ανακαινιστεί το συγκεκριμένο σίνεμα και να μην χτιστούν νέα κτίρια αλλού και χρησιμοποιηθεί μόνο και μόνο για χώρο στάθμευσης. Ελπίζω κάποτε να πάω σινεμά στο πρίσβεν. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε θέματα ίσως όχι τόσο εύκολα. Ευχαριστώ που διευκρινίσατε ότι ο διάλογος για τις βίζες ε, είναι πάντα στο κέντρο των συζητήσεων και των προβλημάτων με το κοσυφοπαίδιο. Έχει αποδειχθεί και εκλογικά ότι το θέμα του κοσυφοπαιδίου νιώθουν ότι απομονώνονται γιατί είναι από τις 15 Δεκεμβρίου είναι η μόνη χώρα που, τις οποίες οι κάτοικοι δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα. Δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω όλα αυτά εδώ, αλλά τα γνωρίζετε. Θεωρούν λοιπόν ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά εις βάρος τους στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έχετε μήπως κάποια ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση στο Συμβούλιο. Χθε είχαμε εδώ τον Βέλγο Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος ε, δυστυχώς είπε ότι είναι κάτι το οποίο ε, θα πρέπει εφόσον δεχτούμε να αλλάξουμε τη θάση μας απέναντι στο κοσφοπέδιο, πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε εσωτερικό επίπεδο και πώς θα γίνει αντιληπτή η αλλαγή αυτής της τάσης από την κοινή γνώμη. Τώρα για τις εκλογές. Ήσασταν ξεκάθαρος λέγοντας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι μια καθαρή κυβέρνηση. Πολλοί φοβούνται ότι θα υπάρξουν για μια ακόμη φορά αρνητικές εκλογικές πρακτικές, θα χρησιμοποιηθούν εκλογικές κάρτες, εκλογικά βιβλιάρια νεκρών, μεταναστών Νομίζω λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει και στα πλαίσια της Επιτροπής Παρατήρησης των Εκλογών να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα. Απαιτείται και οι άλλοι πρέσβοι στην Πρίστινα να διευκρινίσουν ότι ιδιαίτερα εκεί όπου στις εκλογές το 2009 και το 2007 υπήρξαν εκλογικές παραβιάσεις, εκεί θα παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τα πράγματα και εφόσον υπάρξουν απάτες και εφόσον ε, γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν θα εκτιμηθεί σωστά η ψήφος του, τότε αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει να νιώσει ο κόσμος ότι αξίζει τον κόπο να πάει να ψηφίσει σε διάφορες περιοχές. Υπάρχουν ε, επίσης νέοι πολιτικοί οι οποίοι ε, ακριβώς και με τις σύγχρονες απόψεις τους και με εθνικιστικές απόψεις για τη Μεγάλη Αλβανία και τα λοιπά θα κερδίσουν την έδρα τους στις νέες εκλογές και υπάρχει πρόβλημα με τις υπερβολικά εθνικιστικές θέσεις. Αναφερθήκατε επίσης στο θέμα της ε, ενέργειας. Πράγματι η μονάδα παραγωγής εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ε, άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν έχει κλείσει και το πρόγραμμα για τη δημιουργία τρίτου εργοστασίου έχει κολλήσει στην Παγκόσμια Τράπεζα. Υπάρχει ένα θέμα οικολογικό βέβαια, οι μονάδες παραγωγής από άνθρακα ε, ηλεκτρικού ρεύματος εννοώ δεν είναι καλές για το περιβάλλον αλλά σίγουρα θα είναι καλύτερη και νόρια από αυτή που ισχύει σήμερα. Για το EULEX προφανώς υπάρχει εδώ μια ισχυρή παρουσία της Γιούλεξ ακόμα και στον Βορρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια μόνιμη ομάδα της Γιούλεξ που κατοικεί μόνιμα το βόρειο κομμάτι του Κοσμοπεδίου. Και υπάρχουν Σέρβοι στο Βορρά που θέλουν να πάρουν μέρος στις εκλογικές διαδικασίες. Πώς επηρεάζει ο Τάντιτς και η κυβέρνηση των Σέρβων. Εγώ εδώ φοβάμαι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Ευχαριστώ. Κούκαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φάιθ για την ανάλυση που μας παρουσιάσατε για την κατάσταση στο κοσυφοπέδιο. Ήταν δίκαιη και αντικειμενική. Και θα ήθελα επίσης να εκφράσω την εκτίμησή μου για την προσπάθεια που κάνετε εκεί, γιατί η κατάσταση είναι δύσκολη, απαιτητική και υπεύθυνη. Συμφωνώ με τους εισηγητές ότι το βασικό πρόβλημα αυτή την εποχή είναι το θέμα της απελευθέρωσης του συστήματος θεωρήσεων. Όσο νωρίτερα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσει τον διάλογο με αυτούς τόσο το καλύτερο, γιατί κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι οι Κωσοβάροι αυτή τη στιγμή υφίστανται κυρώσεις σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής. Ξέρω ότι το θέμα είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν ε, διαπραγματεύσεις. Όπως έχετε πει, η πολιτική κατάσταση στο Κωσυφοπέδιο είναι πολύ περίπλοκη και ίσως να γίνεται και πιο περίπλοκη με, με τον χρόνο. Υπάρχουν νέα πολιτικά κόμματα, Υπάρχουν κάποιες εσωτερικές εξελίξεις στα παραδοσιακά κόμματα και όλα αυτά καθιστούν την κατάσταση ε, περίπλοκη. Θα είχα πολλές ερωτήσεις να ρωτήσω προς την κατεύθυνση αυτή. Σαν παράδειγμα, η συμμετοχή στις εκλογές. Ακούγονται διάφορα εδώ. Ε, τι πιστεύετε εσείς επί τη βάση και της προεκλογικής εκστρατείας έτσι όπως εξελίσσεται. Η συμμετοχή των Σέρβων τώρα στις εκλογές, η συγγήτρια αναφέρθηκε στο θέμα και εσείς κάνατε κάποια σχόλια. Μπορείτε να μας πείτε κάποια περισσότερα πράγματα, πώς βλέπετε εσείς το μέλλον την συμμετοχή των Σέρβων στις εκλογές. Και μία επιπλέον ερώτηση την οποία δεν ξέρω να διατυπώσω σωστά. Θα το πω λίγο ε, βίαια θα έλεγα. Καλύτερο είναι όμως να τίθεται τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, πράγματι εκτιμούμε τις προσπάθειες που γίνονται σε διπλωματικό επίπεδο. Θα υπάρξει και μια μικρή αντιπροσωπεία θα έλεγα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά θα υπάρξει έλλειψη παραδοσιακών εκλογικών ε, ε, αποστολών Και μήπως πιστεύετε ότι το αλβανικό σενάριο θα επαναληφθεί και στο κοσυφοπέδιο. Ξέρουμε τι γίνεται στην Αλβανία, ξέρουμε ποια είναι η δυσκολία και πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια τέτοια κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σας ότι μετά τις εκλογές το κοσυφοπέδιο έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση η οποία θα συγκεντρώσει την προσοχή της στην δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα Τέτοιου είδους λοιπόν πολιτικοί καυγάδες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση θα κάνουν ε, πολύ πιο ε, δύσκολη την κατάσταση. Ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται και νομικά θέματα αμέσως μετά τα ε, αποτελέσματα ενώ θα πρέπει ε, η κυβέρνηση να ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση της χώρας, να βρει μια λύση για τους ανέργους και όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν κάποια πρόταση σχετικά με την ε, αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης. Και εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, ο κ. Προβέρα σχετικά με την κατάσταση του νόμου και της τάξης στη χώρα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ, μεγα... πολύ σημαντικό πολύ σημαντική η επίπτωση της εγκληματικότητας στις διάφορες, ε, στα διάφορα στρώματα της κοινωνίας, όχι μόνο του κοσφοπεδίου. Εμπλέκεται η εγκληματικότητα και στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, στην οικονομία, και γενικά σε συμπεριφορές οι οποίες είναι παραβατικές και απαράδεκτες. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν. Και μια τελευταία ερώτηση. Η στάση της σερβικής μειονότητας, κοινότητας. Υπήρξε συμμετοχή και όπου όχι, πού ήταν τα προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Φάιτ που είστε εδώ. Δείξατε σωστά πώς έχει η κατάσταση, αν και βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω πια αμφιβολίες για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. οι διαδικασίες βελτίωσης των πραγμάτων είναι πάρα πολύ αργές και σε επίπεδο κοινωνικό και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο κράτους διεκαίου και σε επίπεδο εγκληματικότητας και σε επίπεδο σεβασμού του διαχωρισμού των εξουσιών και σε σχέση με την κατάσταση στη Μητρόβιτσα. Γενικά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι και η κοινή γνώμη του κοσμοπεδίου βλέπει με διαφορετικό τρόπο την Ευρώπη. Ακολουθούν θα έλεγα μία μορφή έτσι απόκριφου φετιχισμού σε σχέση με κάποιες βασικές αρχές που τους οδηγεί σε απαράδεκτες εκφάνσεις εθνικιστικές. και από πλευράς μας υπάρχει μια αντιφατική θα έλεγα πολιτική και μια αντιφατική στάση. Σε όλες τις εκθέσεις που έχουμε κάνει και παρόλες προσπάθειες που έχουμε κάνει, πέντε χώρες δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του κοσυφό πεδίου. Υπάρχει το θέμα βέβαια της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων, από την άλλη ε, δεν είναι μόνο εκεί το θέμα, υπάρχουν θέματα πολιτικά πραγματικά που χρήζουν προσοχής. Δεν ξέρω αν είστε κι εσείς τόσο σκεπτικιστής όσο εγώ, δεν είναι απαραίτητο βέβαια. Να σας θέσω τώρα κάποιες ερωτήσεις. Ανάμεσα στους θετικούς στόχους, τους οποίους επιδιώκει η κυρία Άστον και που δεν είναι και πάρα πολύ κατάφερε να ξαναφέρει σε επαφή τις αρχές του Κοσφοπεδίου με τις αρχές της Σαρβίας. Αυτές οι επαφές είναι χρήσιμες βέβαια για τη χώρα. Υπάρχει όμως μια αντίληψη η οποία ενισχύεται ότι η Σερβία ανεξαρτήτως του μελόντος του κοσυφοπεδίου θα μπορούσε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το κοσυφοπέδιο. Δεν ξέρω αν ακούγεται αυτή η συζήτηση και ε, στο κοσυφοπέδιο και αν ναι, αν δημιουργεί προβλήματα για την πρόοδο της κατάστασης. Δεύτερη ερώτηση. Πριν λίγο καιρό είχα πάει στο Κωσυφοπέδιο στις κοινοτικέ εκλογές και μου έδειξε η επίσκεψη αυτή ότι είχαμε πάντα ένα πρόβλημα για να συνδυάσουμε όλους τους πρωταγωνιστές της περίπτωσης της συγκεκριμένης, δηλαδή αναπτυξιακή συνεργασία, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, Υπάρχει έλλειψη συντονισμού δηλαδή και απαιτείται να υπάρξει περισσότερο συντονισμός. Και τέλος, θα ήθελα την άποψή σας εάν πράγματι από αυτές τις πολιτικές εκλογές, οι οποίες θα ελπίζω να γίνουν με μεγάλη διαφάνεια, μπορεί να αποσταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την υπευθυνοποίηση των πολιτικών δυνάμεων που συμμετέχουν στις εκλογές αυτές. Καλώς. Τελευταία Ομιλία Λίζεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Πρέσβη για την πολύ εμπεριστατωμένη και μεστή παρουσίαση και με ιδιαίτερη χαρά άκουσα κάποιων επαΐων, επαΐων τα πραγματικά του θέματος. Θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις για οικονομικά ζητήματα. Μιλήσατε για τις ε, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις του Κωσυφοπεδίου με τις γειτονικές χώρες. Μιλήσαμε για τις, χώρες με, για τις σχέσεις με τη Σερβία που είναι για ευνόητους λόγους κάπως δυσχερείς, με τις υπόλοιπες όμως χώρες ε, ε, της γειτονίας του. Με την Αλβανία, για παράδειγμα, τι σχέσεις έχει το Κωσυφοπέδιο, πολιτικές και οικονομικές. Και πάλι για οικονομικά θέματα. Μιλήσατε για την οικονομική κατάσταση στο Κωσυφοπαίδιο που είπατε ότι είναι αρκετά ζωφερή και απεσιόδοξη και μιλήσατε για την ανάγκη επενδύσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω γιατί πρόσφατα ε, μίλησα με κάποιον αξιωματούχο της αστυνομίας που πέρασε, της Πολωνίας που πέρασε αρκετά χρόνια στο Κωσυφοπαίδιο. Πώς ε, πώς μπορεί να διαβιώσει το κοσυφοπέδιο, τι πλούτο έχει, τι έσοδο μπορεί να έχει για τον προϋπολογισμό, σε ποιον οικονομικό κλάδο πιστεύετε ότι θα μπορέσει να στηριχθεί για την οικονομική του ανάπτυξη το κοσυφοπέδιο. Και ο κύριος Στάνοκ ήρθε στο μεταξύ και ζητάει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ειδικέντο Ταλμένα, Πρόσφατα και εγώ πήγα στο Κωσυφοπαίδιο και συμμερίζομαι τις ανησυχίες των συναδέλφων και μάλιστα την κατάσταση την είχα προβλέψει αρκετά πριν. Άλλο θέμα όμως αυτό. Έχω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Γιατί είμαι ο εισηγητής για το Μαυροβούνιο, αλλά ισχύει και για άλλες ε, χώρες. Και στο Κωσυφοπέδιο έχουμε εσωτερικά εκτοπιστέντες από τις κοινότητες Ρωμά, Ασκάλη και Αιγυπτιακή τι κινήσεις κάνετε και τι πίστα ασκήσετε στην κυβέρνηση προκειμένου να μπορέσουν οι κοινότητες αυτές να επαναπατριστούν, να γυρίσουν στα σπίτια τους στο κοσυφοπαίδιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα να γυρίσουν πολύ Σέρβοι, αλλά οι άλλε κοινότητε θα ήθελαν να γυρίσουν. Τι συγκεκριμένα προσπάθειε γίνονται για αυτέ τι τρει κοινότητε στο Κωσυφοπαίδιο, Ρωμά, Ασκάλη και Αιγυπτιακή. Δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο, οπότε θα σας δώσω το λόγο κύριε Πρέσβη για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές, τα μέλη της Επιτροπής, για τις ερωτήσεις που έθεσαν και την γενική υποστήριξη που μου παρήχαν. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου με βάση τα κεφάλαια που σας παρουσίασα και στην αρχική μου εισήγηση. Πολλές ερωτήσεις τέθηκαν για τις επερχόμενες εκλογές. Με ρωτήσατε τι προετοιμασία γίνεται, πώς θα διεξαχθούν και ποια είναι η πιθανή έκβαση αυτών των εκλογών. Επίσης με ρωτήσατε τι θα γίνει με την μετεκλογική κατάσταση. Δηλαδή ποιες θα είναι οι πολιτικές, οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Θα απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις για οικονομικά θέματα και για τις θεωρήσεις. Αυτά θα είναι τα τρία βασικά κεφάλαια. Θα ήθελα να σας πω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στείλουμε το μήνυμα ότι θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς ίσομη η παγκόσμια κοινότητα αυτές τις εκλογές. Και όταν λέω εμείς θα παρακολουθήσουμε, ενώ ότι συνεργαζόμαστε στενά και με τις Ηνωμένε Πολιτείε που ε, επιδεψιλεύουν πόρους στις ομάδες της οργανώσεις παρατήρησης εκλογών. Και φυσικά θα έχουμε και συνεργασία και με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, υπό τον τίτλο «Δημοκρατία και δράση». Συντονισμένες λοιπόν δράσεις θα έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους Αμερικανούς που θα φέρουν περίπου 5.000 ανθρώπους στα εκλογικά κέντρα για να παρατηρήσουν τη διεξαγωγή των εκλογών. Και δεν θα παρατηρήσουμε μόνο την κατάσταση στα εκλογικά κέντρα, θα εξετάσουμε και το θέμα της μεταφοράς των καλπών και θα είμαστε παρόντες και στο κέντρο καταμέτρησης των ψήφων. Επίσης θα εξετάσουμε και διάφορες διαδικασίες προσφυγής ή αιτιάσεων παραπώνων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έστειλε ήδη τρεις εμπειρογνώμονες που ήδη προβαίνουν σε μια προκαταρκτική ανάλυση για τον τρόπο προετοιμασίας των εκλογών. Εξετάζουν το κατά πόσο το νομικό πλαίσιο είναι σωστό. Και η πρώτη εντύπωση που αποκόμισα από τους εμπειρογνώμονες αυτούς είναι ότι η γενική τους αξιολόγηση είναι θετική. Θα ήθελα όμως να επισημάνω ότι το Μητρό Ψηφοφόρων, οι κατάλογοι των ψηφοφόρων δεν είναι ενημερωμένοι. Εν μέρει γιατί ε, οι εκλογές διοργανώθηκαν πολύ γρήγορα. Η αναγγελία για τις εκλογές έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και αποτέλεσμα θα είναι ότι η προσέλευση στις κάλπες θα είναι υψηλότερο από τις στατιστικές προβλέψεις. Γιατί πολλοί που πέθαναν έχουν ε, αφαιρεθεί από τους εκλογικούς καταλόγους. Αλλά και πάλι οι εκλογικοί κατάλογοι δεν μας δίνουν μια ακριβή εικόνα γιατί είναι πολύ περισσότεροι ε, αυτοί που ζουν και έχουν επιστρέψει στο κοσυφοπέδιο. Αλλά δεν ξέρουμε αν η προσέλευση θα φτάσει στο 50% ή θα είναι και υψηλότερη. Θα εξαρτηθεί, θα εξαρτηθεί και από τις καιρικέ συνθήκες το πόσοι ψηφοφόροι θα πάνε να ψηφίσουν. Πάντως, σε ό,τι αφορά την ψήφα των Σέρβων, εκεί περιμένουμε όντως άθρα ε, προσέλευση και ελπίζω να φτάσουμε στο ίδιο ποσοστό προσέλευσης ε, με αυτό των πρόσφατων δημοτικών εκλογών. Και άρα μεγαλύτερο ποσοστό προσέλευση από ό,τι στις γενικές εκλογές του 2007, τις βουλευτικές. Σε ό,τι αφορά την ψήφο των Σέρβων στο Βορρά και την προσέλευση του Κάλπες, θα ήθελα να πω ότι Λυπάμαι που ε, η έκκληση για μποϊκοτάρισμα απευθύνθηκε από, τους, ε, τις παράλληλες αυτές δομές και δημάρχους του Βορρά. Πραγματικά αυτό είναι αντιπαραγωγικό γιατί δεν συνάδει με τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαντάζομαι, ελπίζω να συμφωνείτε κι εσείς με αυτό. Και η δήλωση του Προέδρου Τάντιτς στη διάσκεψη κορυφής της ΟΑΣΕ ότι οποιαδήποτε αλλαγή επιτόπου θα σημάνει το τέλος του διαλόγου με την Πρίστινα, μας κατέβλεξε κάπως αυτή η δήλωση, γιατί η πραγματικότητα επιτόπου και η κατάσταση επιτόπου καθορίζεται από τους πολίτες και όχι από τις κυβερνήσεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Και νομίζω θα πρέπει να είναι σαφής εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν οι πολίτες ζητούν δημοκρατικές αλλαγές και στο βόρειο κοσυφοπαίδιο, αν αυτή είναι η λαϊκή τιμιγορία, δεν νομίζω ότι καμία κυβέρνηση δικαιούται να εμποδίσει την ικανοποίηση αυτή τη λαϊκή βούληση. Ελπίζω να συμφωνείτε. Οπότε θα έχουμε ίσω κάποια απογοήτευση στο βόρειο Κόσοβο. Και με το πλαίσιο που επικρατεί στο βορρά γνωρίζω ότι κάποιοι θα προτιμούσαν να, ακόμη και να ιδρύσουν ένα νέο πολιτικό κόμμα. Ο ηγέτης του μάλιστα ε, δέχτηκε τριπλή επίθεση με χειροβομβίδες ε, στην, στο σπίτι του και δέχτηκε επιθέσεις και η οικογένειά του. Αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει η κατάσταση αυτή οπωσδήποτε να αλλάξει. Δεν θα πρέπει φυσικά να υπάρξει γνωθεία, αλλά ούτε και δηλώσεις των πολιτικών ηγετών της αλβανοκοσοβάρικης κοινότητας που προβλέπουν την έκβαση των εκλογών πριν ακόμη γίνουν, γιατί δημιουργούνται κακές προϋποθέσεις, δυσπιστία, δυσάρεστο κλίμα και ίσως αυτά μας τρέψουν προς λάθος κατεύθυνση. Και κάποιοι πολιτικοί που κάνουν υποσχέσεις που γνωρίζουν κάλλιστα ότι αποκλείεται να τις στηρίσουν. Να τις, μιλούν για αυξήσει μισθών της τάξης του 30 και 50%. Φυσικά είναι ευκταίο κάτι τέτοιο, αλλά είναι ανέφικτο. Ιδιαίτερα για έναν προϋπολογισμό μιας χώρας σαν το Κόσοβο. Σε γενικές γραμμές λοιπόν, Σε ό,τι αφορά την προετοιμασία των εκλογών, έχουμε μπει στο δρόμο αυτό προς εκλογές και μέχρι στιγμής δεν έχουμε ενδείξεις για παρατυπίες και ατασταλίες στη διεξαγωγή των εκλογών. Το δεύτερο σημαντικό κόμμα στο Κωσυφοπέδιο, το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα, το LDK, έχει ανακτήσει με την ηγεσία ένα τμήμα της υποστήριξης των ψηφοφόρων. Οπότε στην προεκλογική εκστρατεία ε, υπάρχει σχετικά ισοτιμία μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι αρνητικά τα αποτελέσματα των εκλογών. Και μετά την εμπειρία που είχαμε με τις δημοτικές εκλογές, πιστεύω ότι οι τελευταίες εκλογές θα ανταποκρίνονται στις υψηλές διεθνείς προδιαγραφές και ελπίζω ότι και η αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει να προβεί σε μια σαφή αξιολόγηση αμέσως μετά την διεξαγωγή και την καταμέτρηση. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε κάποιους τομείς που θα απασχολήσουν τη νέα κυβέρνηση και ιδιαίτερα να αναφερθώ σε κάποια οικονομικά ζητήματα. Πιστεύω ότι η οικονομία θα πρέπει να λάβει υπόψη τα συγκριτικά αποτελέσματα και το δυναμικό του, γιατί το Κόσοβο έχει πολλούς νέους, πρόθυμους, εργατικούς, που είναι, πρόθυμοι, είναι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με σχετικά χαμηλούς μισθούς, έχει φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα ρηκτό πλούτο η γεωγραφική θέση του, τοποθεσία του Κωσυφοπεδίου είναι επίσης προνομιακή. Βρίσκεται στο κέντρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Βρίσκεται στην καρδιά αυτής της περιοχής. Υπάρχουν τέτοια συγκριτικά πλεονεκτήματα που μπορεί να αξιοποιήσει το Κωσυφοπέδιο για να μεγεθύνει την οικονομία του και να φτάσει σε επίπεδα εφάμιλα με άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Φυσικά η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα. Περιμένουμε την διεκπαιρέωση της ε, ιδιωτικοποίησης του ηλεκτρισμού, της παραγωγής ενέργειας και φυσικά περιμένουμε να δούμε και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της συνέχειας ε, λειτουργίας του εργοστασίου, ενός εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να κλείσει τα επόμενα χρόνια και περιμένουμε να συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα με μια πρόταση για κατασκευή ενός νέου ηλεκτρικού σταθμού που θα λέγεται Κόσοβο Γ και θα αντικαταστήσει τον Κόσοβο Α που θα κλείσει. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Σα μίλησα για τις σχέσεις του Κωσυφοπεδίου με τη Σερβία. Σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Αλβανία, όπως φαντάζεστε, οι σχέσεις Κωσόβου και Αλβανίας είναι στενές και σε οικονομικά θέματα. Η Αλβανία είναι σημαντικό εταίρος του Κωσυφοπεδίου και υποστηρίζει το Κωσυφοπέδιο σε πολλούς τομείς και τις πολιτικέ προσπάθειες του Κωσυφοπεδίου για να τύχει όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση από την παγκόσμια κοινότητα. Και Υπάρχουν και εμπορικοί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών. Πολλές φορές δυστυχώς αυτοί οι δεσμοί είναι παράνομοι και γίνονται επιχειρήσεις που καλό θα ήταν να, να μην παίρνουν απαρατήρητες γιατί υπάρχει και διακίνηση, υποπτή διακίνηση προσώπων και υπάρχει δυνατότητα έκδοσης αλβανικών διαβατηρίων για Κωσοβάρους. Αυτό είναι ενδιαφέρον ζήτημα υπό το πρίσμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Συμφωνώ και όσοι μερίζομαι τις ανησυχίες του κυρίου Παντζέρη και της δικές σας κύριε Πρόεδρε ως προς τα υψηλά επίπεδα διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Πάντως, δεν θα πρέπει να τραγικοποιούμε τα πράγματα. Αυτό το φαινόμενο δεν είναι ίδιο του κοσυφοπεδίου μόνο. Δυστυχώς είναι γενικό φαινόμενο στην περιοχή. Έχουμε μια αποστολή πάντως κράτους δικαίου με γύρω στα 2.000 άτομα προσωπικό που ελέγχει καθημερινά και προσφέρει συμβουλές ε, στην αστυνομία, στο δικαστικό σύστημα και παρακολουθεί γενικώ την κατάσταση στα θέματα αυτά και σίγουρα θα πρέπει κατεπηγόντω να ενισχυθεί ο δικαστικό κλάδο, αλλά πρόοδο υπάρχει και είναι τεράστια η επένδυση που έχει κάνει στον τομέα αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκεί να στυλιτεύουμε ή να διτυμπανίζουμε τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες των ε, θεσμικών οργάνων του κοσυφοπεδίου, ενώ γνωρίζουμε ότι ταυτόχρονα επενδύουμε ε, πάρα πολλά στη χώρα αυτή. Έχουμε τη μεγαλύτερη αποστολή, τη ULEX στο Κωσυφοπαίδιο, μη στρατιωτική. Και πιέζουμε για περισσότερα αποτελέσματα, για εντατικοποίηση των ερευνών και των διώξεων των εγκληματιών και επίσης ζητούμε δραστηριοποίηση ορατότητα και παρουσία της Γιούλεξ στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Και εγώ είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη ότι αφορά τα... τις ενέργειες που κάνει η Γιούλεξ προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά υπάρχει και ένας ευρωσκεπτικισμός στο Κωσυφοπαίδιο, είναι συνέπεια όλων όσων προαναφέραμε, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω ότι αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκε η, η μείωση της υποστήριξης για την ένταξη του κοσμοπεδίου έχει μειωθεί στο 10% αλλά έχει μειωθεί κατά 10% δηλαδή το 75% υποστήριξη έχουμε 65% δεν είναι τραγικά τα πράγματα δηλαδή αλλά προτιμούμε να μην συνεχίσει αυτή η ευθύνουσα πορεία σε ό,τι αφορά την ε, υποστήριξη του λαού για την ένταξη του κοσμοπεδίου σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, μην με παρεξηγήσετε, αλλά δεν πρόκειται να κάνω δηλώσεις που μπαίνουν στα χωράφια αρμόδιων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι το θέμα είναι πολύ λεπτό, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει είναι να είμαστε συνεπείς στα μηνύματά μας να μην ε, έχουμε αντιφατικά μηνύματα από τους επιτρόπους. Να μην λέει τη μια μέρα ο υπουργό Εξωτερικών ε, ε, μιας χώρας το α και την άλλη μέρα ο υπουργό Εξωτερικών της ίδιας χώρας να λέει κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να αποφύγουμε τις αντιφάσεις. Αλλά η ευρωπαϊκή προοπτική δεν είναι μια αυτόματη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό το έχουν καταλάβει όλες οι χώρες της περιοχής. Αλλά δημιουργεί μία αβεβαιότητα αυτή η αντιφατικότητα. Και αυτό επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη που επικρατεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις χώρες αυτές. Κύριε Τάνοκ, έρχομαι στην τελευταία μου παρατήρηση. Έφυγε στο μεταξύ ο κύριος Τάνοκ. Ρώτησε όμως για τη θέση των ε, τριών κοινοτήτων Ρωμά, Ασκαλή και Αιγυπτίων. προσπαθούμε να εφαρμόσουμε κάποια αναπτυξιακά προγράμματα για επαναπατρισμένους που καλύπτουν και τις κοινότητες αυτές. Νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία πια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί τα θεσμικά όργανα του Κωσυφοπεδίου πια πληρούν τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνονται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως η όλη διαδικασία της παλινόστησης ή του υποχρεωτικού επαναπετρισμού είναι επώδυνη και δυσχερής γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες στην οικονομία για τους παλινοστούντες και οι Ρωμά ιδιαίτερα βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη κατάσταση. Πάντως το μήνυμα που εγώ θα ήθελα να στείλουμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ ως ειδικό συντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επαφές που θα έχω με, άλλες, με άλλους απεσταλμένους και ειδικού συντεταλμένους όπως τον ομολογό μου των Ηνωμένων Πολιτειών παρακολουθούμε τα πράγματα και τις εξελίξεις καθημερινά παρέχουμε συμβουλές και μεριμνούμε για την ε, τήρηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των διαφόρων κοινοτήτων. Και όσο θα συνεχίζεται η εντολή μου, εγώ θα δώσω ιδιαίτερη έφαση στο θέμα αυτό των μειονοτήτων. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία σας και εμπεριστατωμένη. Σας περιμένουμε και την επόμενη φορά για ενημέρωση ως προς τις τελευταίες εξελίξεις. Ευχαριστώ.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 Έκθεση Μακοβέη για την έκθεση παρατήρησης των εκλογών στη Μολδαβία. της 28 Οκτωβρίου. Διεξήχθησαν ειρηνικά οι εκλογές αυτές σε ένα πλουραλιστικό κλίμα και σύμφωνα με τα επίπεδα τα ευρωπαϊκά πάνω κάτω. προείδρευε της αποστολής η κυρία Μακοβέη, η οποία θα μεταφέρει τα συμπεράσματα της επίσκεψής της. Έχετε το λόγο κυρία Μακοβέη. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν, 28 Νοεμβρίου, παρακολουθήσαμε τις εκλογές ε, στην Μολδαβία, όπω είπατε, ήμασταν τέσσερις, τέσσερα βουλευτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφου που ήρθαν μαζί μου και να ευχαριστήσω και τη γραμματεία για την ενίσχυση κάτω από σημαντική πίεση χρόνου. Είχαμε σε 31 εκλογικά, 31 εκλογικά κέντρα, στην Κακαούτσια, στην Ίστρα, παντού θα ήθελα να σας πω ποιες ήταν τα αποτελέσματα, τα τακτικές, επαγγελματικέ διαφανείς και δίκαιες οι εκλογές αυτές. Είδαμε να υπάρχει σημαντική πρόοδος από την περασμένη φορά. Τα, η τηλεόραση και η ραδιοφωνία, η παρουσίαση ήταν πολύ δίκαια. Η επιτροπή ήταν επίσης ε, επαγγελματική. Επίσης, είδαμε μια καλή εκστρατεία να προσκληθούν όλοι να ψηφίσουν, Ακόμα και οι επιστολές που τους έστελαν στα σπίτια τους, τους είπαν με τη διεύθυνση, εκεί θα πρέπει να πάνε να ψηφίσετε μεταξύ αυτής και αυτής της ώρας. Επίσης ηλεκτρονική καταγραφή των εκλογέων ένα σύστημα που επελέχθη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκε από το Ηνωμένα Έθνη και το είδαμε εν λειτουργία την ημέρα των εκλογών. 60% ήταν η συμμετοχή στι εκλογέ είναι πολύ υψηλό το ποσοστό αυτό, δεδομένου ότι στου 18 τελευταίου μήνε έλαβε χώρα τρεις ε, κοινοβουλευτικέ εκλογέ. και επίση θα ήθελα να σου πω ότι 60.000 ε, άτομα περίπου ψήφισαν από το εξωτερικό. 20 ε, κόμματα υπήρχαν και 19 ανεξάρτητοι ε, υποψήφοι, 39 δηλαδή σε σύνολο. Το εκλογικό δελτίο είχε μήκο ένα μέτρο. Οι ερασαλίες ήταν πάρα πολύ λίγες, μεμονωμένες και οπωσδήποτε έχει περισσότερες από τις άλλες χώρες. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να πω. Οι διαπραγματεύσει για τα πρώτα προσωρινά αποτελέσματα και συμπεράσματα με τη βοήθεια του κυρίου Τονίνου Πισούλη, επικεφαλή τη αντιπροσωπείας και τον κύριο Ιντρεξάρ που ήταν ο εκπρόσωπος, ο επικεφαλής της, της αντιπροσωπείας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεργασία με τις άλλες αυτές αντιπροσωπείς ήταν κάπω δύσκολη. Καταφέραμε όμω τελικά να καταλήξουμε σε μια κοινή δήλωση. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ότι η διαφωνία αυτή λόγω της αλλαγή στον εκλογικό νόμο που έγινε το καλοκαίρι του 2010. Το κατόφλιο μειώθηκε από το 5 στα 4% ε, οι φοιτητέ ε, είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ε, εκεί που σπουδάζουν, γιατί ορισμένοι θα είχαν προλάβει να πάνε στις πόλεις από που κατάγοντο. Επίσης το σύστημα από αναλογικό μετατράπηκε σε ένα σύστημα ίσης κατανομής, δηλαδή όλες οι εκλογές και οι εντολές εκείνων που δεν έφτασαν στο 4% καταμερίστηκαν επίσης όρις σε, σε, στα άλλα κόμματα ή στους υποψηφίους που πέρασαν. Αυτό είναι υπέρ της, των μικρών κομμάτων βέβαια, είτε στην αντιπολίτευση της κυβέρνησης, αλλά οπωσδήποτε είναι ε, μια μέθοδος που επελέχθη πότε έγινε, που, που, που έγινε η διαφωνία, γιατί η Επιτροπή για τις καλές πρακτικές ε, προβλέπει μία παράγραφο για το θέμα αυτό που λέει ότι οι αλλαγές του εκλογικού νόμου δεν θα πρέπει να γίνονται ε, συντομότερα προς εκλογές από ένα έτος. Τώρα βέβαια εδώ έχουμε μια πολιτική κρίση και ε, ανάγκη επίγουσας ε, αλλαγής της κυβέρνησης. Και θα έλεγα ότι όταν έχουμε σε 1,5 χρόνο τρεις εκλογές και ένα δημοψήφισμα επιπλέον και το θέμα της πολιτικής κρίσης, έχουμε μια έκτακτη κατάσταση. Και θα πρέπει ο να ανταποκριθεί στην πολιτική κρίση. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, δεν είναι πια εδώ πολλοί συνάδελφοι, αλλά ας πω να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης απέστειλε δύο επιστολές πριν από μερικούς μήνες και που λένε ότι αυτές οι αλλαγές είναι σύμφωνες με την ευρωπαϊκή κληρονομιά στον τομέα των εκλογικών νόμων και δεν θα παρεμποδίσουν τις ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Δηλαδή το Συμβούλιο της Ευρώπης είπε κατά βάση ότι εντάξει οι ελεγές αυτές. Και γι' αυτό μου φαίνει και περίεργο ε, η στάση αυτή των ε, συναδέλφων από τις άλλες ε, κοινοβουλευτικές εκπροσωπήσεις που στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας είπανε ότι θα πρέπει να δώσουμε κάποια επιχειρήματα στο Κομμουνιστικό Κόμμα να διαμαρτυρηθεί κατά των αποτελεσμάτων, αν το αποτελεσμάτων θα πρέπει. Δεν ήταν αυτός ο ρόλος μας όμως να είμαστε εκεί. Και επαναλαμβάνω, καταλήξαμε σε ένα συμβαστικό κείμενο. Βλέπετε ότι είναι ισορροπημένο. Όλες οι απόψεις παρουσιάζονται. Και θα περάσω τώρα στο τρίτο τμήμα, ίσω το πιο ενδιαφέρον και το πιο σημαντικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών και αυτό τι σημαίνει. Λοιπόν, τα αποτελέσματα των εκλογών ήταν ότι έχουμε 101 έδρε, το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε 42 έδρες και όλοι οι άλλοι φιλελεύθεροι δημοκράτες κλπ. Είναι τώρα σε, με 59 ε, 59 έδρες, ένας ε, ένα σεισμός υπέρ της ε, Ευρώπης. Έχουν την πλειοψηφία, αλλά δεν αρκεί η πλειοψηφία αυτή για να πετύχουν την εκλογή του Προέδρου, γιατί για την εκλογή του Προέδρου σύμφωνα με την ε, νομοθεσία της χώρας έως 61 ψήφου, ψήφοι, λείπουν δηλαδή δύο, και γι' αυτό γίνονται τώρα μια σειρά διαπραγματεύσεων. Δεν θα μπορεί μια χώρα να επιβιώσει χωρίς Πρόεδρο. Χωρίς να αντικαταστήσει δηλαδή τον Πρόεδρο. Ένας πρόεδρος χρειάζεται βέβαια γιατί ακριβώ το Σύνταγμα προβλέπει ότι αν δύο φορές θα πετύχει στην ε, εκλογή του Προέδρου η Βουλή θα ξαναγίνουν κοινοβουλευτικέ εκλογές και αυτό δεν το θέλει κανένας, θέλει να υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση που να υιοθετήσει κάποια μέτρα προ όφελο τη χώρα και προς την δημοκρατία. Άστον Φίλε, ο Αμερικανός πρέσβους, έκαναν διάφορες δηλώσεις. Όλοι είναι πρόθυμοι και ανοιχτοί να βοηθήσουν στη δημιουργία κυβέρνησης. Και εγώ θα σας κρατήσω ενημερούς για τις εξελέξεις και για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Αντρική ναι, έχετε το λόγο. Οι εκλογές λοιπόν που έγιναν στην Μολδαβία την προηγούμενη Κυριακή ήταν οι πρώτες εκλογές τις οποίες μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε. Από την άλλη ήταν η τρίτη φορά ε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε μπορέσει να είναι παρόν μπορώ να καταλήξω σε ορισμένα συμπεράσματα. Ε, νομίζω ότι οι εκλογές ήταν βασικά δημοκρατικές. Οι εκλογές σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να γίνονται ε, με τα ίδια στάνταρτς και αυτό έγινε και στη Μολδαβία. Νομίζω ότι είχαν οργανωθεί σωστά και η καταμέτρηση είχε οργανωθεί σωστά Υπήρχαν 10 ε, παρατηρητές περίπου σε κάθε εκλογικό κέντρο και νομίζω ότι μπόρεσαν να παρατηρήσουν σωστά τις εκλογές. Το 60% των εκλογέων πήραν μέρος στις εκλογές υπήρξε η δυνατότητα ε, της προεκλογικής εκστρατείας, της διεξαγωγής της προεκλογικής εκστρατείας α, ικανοποιητική. Και θυμίζω ότι ανάμεσα στους παρατηρητές υπήρχαν και 600 διεθνείς παρατηρητές. Από το Κοινοβούλιο ήταν μόνο τέσσερις. Νομίζω ότι η προσοχή που δώσαμε στη Μολδαβία δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έστειλε 30 παρατηρητές. Υπήρξαν βέβαια μεμονωμένοι παρατηρητές από τα κράτη-μέλη, αλλά έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει περισσότερο κόσμο, λαμβάνοντας υπόψη τα προγράμματα τα οποία εμείς ε, εφαρμόζουμε στη συγκεκριμένη αυτή χώρα. Από το 2009 η χώρα αυτή θυμίζω ότι δεν είχε παρά μόνο ε, μεταβατικό πρόεδρο και οι εκλογές ήταν απαραίτητες και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μπήκαν στον κόπο να πάνε στη Μολδαβία. Κατά τη διάρκεια των παλαιών αποστολών εκλογικών στη χώρα αυτή είχαμε πει ότι υπήρχαν προβλήματα για τους Μολδαβούς που κατοικούν στο εξωτερικό. Αλλά υπήρξαν εκλογικά κέντρα τώρα σε 13 χώρες εκτός Μολδαβίας για να μπορέσουν να ψηφίσουν και χρησιμοποιήθηκε. 28.000 Μολδαβοί ψήφισαν στην Ιταλία, στη Ρουμανία, στην Ισπανία, στη Ρωσία και τα λοιπά. Στην Πάντοβα, στο Παρίσι, στη Μόσχα τέλειωσαν και τα ψηφοδέλτια. Ε, κανένας δεν πίστευε ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον των Μολδαβών του εξωτερικού για την εκλογική διαδικασία. Για την κατάσταση τώρα μετά τις εκλογές υπήρξε αναφορά στις έδρες από τον αρχηγό της ε, Επιτροπής Παρατήρησης. Υπάρχει δυνατότητα να καταλήξουν σε μια κάποια συμφωνία τα τέσσερα κόμματα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η συμφωνία αυτή, αλλά πάντως Υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας και με το Κομμουνιστικό Κόμμα και όλα τα πολιτικά κόμματα γενικά προσπαθούν να περάσουν σε, μια, σε έναν επικοδομητικό ε, συμβιβασμό και η αντιπολίτευση θα πρέπει και αυτή να είναι επικοδομητική και να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της χώρας στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ πρέπει του χρόνου να επισκεφθεί τη Μολδαβία και αυτό θα επηρεάσει θετικά τη χώρα και τις προσπάθειες της χώρας αυτής να καταλήξει σε μια επίλυση των προβλημάτων της. Οι Μολδαβοί αξίζουν την απαραίτητη σταθερότητα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπε ότι ε, δεν θα κάνει κανονική παρέμβαση αλλά θα συνεργαστεί με την κυβέρνηση της χώρας και η κυβέρνηση πρέπει να είναι σταθερή για να αναλάβει τις ευθύνες της. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γουότσον. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μακοβέη για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και να τη συγχαρώ για την προσπάθεια που έχει κάνει εξ ονόματος του Κοινοβουλίου. Η κυρία Ένε είπε ότι δεν ήταν μεγάλη αντιπροσωπεία, πράγματι δεν ήταν μεγάλη, αλλά ποιοτικά ήταν πολύ σημαντική. Θα ήθελα να συγχαρώ και την Μολδαβική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή μιας εκλογικής διαδικασίας επιτυχούς. Θα ήθελα επίσης ε, να ε, συμμετέχω και ε, στις εορτές και όχι ε, και στις γενικότερα μπορεί να διαφωνεί κανείς με τις επιλογές αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το κόμμα που υποστηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αύξησε τον αριθμό των θέσεων των εδρών στη Βουλή, οι κομμουνιστές έχασαν θέσεις και υπάρχει μια ξεκάθαρη εντολή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και τη συνέχισή της. Προσωπικά λυπάμαι βέβαια κάποιες δηλώσεις που ακούσαμε από τον Επίτροπο Φούλε και την, Επίτροπο... και την Βαρόνη Άστον. Δεν υπήρξε πλήρης αναγνώριση του συγκεκριμένου γεγονότος και του πώς θα συνεχιστούν τα πράγματα. Κατανοώ την δυσφορία των ηγετών των δημοκρατικών κομμάτων με την κατάσταση στην οποία έχουν περιπέσει πλέον. Μια κατάσταση η οποία δεν θα τους επιτρέψει να επιλέξουν πάλι πρόεδρο μάλλον. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι το μήνυμα το οποίο θα πρέπει να σταλεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω οποιασδήποτε ρύθμιση συνεργασίας με τους κομμουνιστές και με τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον κύριο Φιλάτη από ποιον άλλο πολιτικό είναι ένα μήνυμα το οποίο θα τύχει μάλλον ψυχρής απάντησης. Πολλοί από εμά έχουμε ανησυχήσει γιατί η διαδικασία το να φέρουμε κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις χώρες ε, ε, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, εννοώ τις χώρες γειτονίας, είναι μια διαδικασία που απέτυχε. Τα πράγματα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν άλλη προοπτική και να ενισχυθούν οι θέσεις που έχουμε εμείς. Φαίνεται ότι η Ένωση δεν έχει μειώσει όμως την επιρροή της στις χώρες αυτής, αυτής της κατηγορίας. Η αντιπολίτευση ισχυροποιείται, εν πάση περιπτώσει, και το μήνυμα που στέλνουμε στη Μολδαβία είναι ότι θάψτε τις εσωτερικές σας διαφορές και δουλέψτε για την πρόοδο της χώρας σας και να δούμε αν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή και με τον Προεδρεύοντα. Και να πούμε επίσης στην, στο κόμμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κάντε περαιτέρω προσπάθειες για να πετύχετε μεγαλύτερη υποστήριξη και αν χρειαστεί ξανακάνετε εκλογές και πάρτε πιο ξεκάθαρη εντολή από το λαό. Λοιπόν, ε, εξ ονόματος της ομάδας μου η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στην αντιπροσωπεία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους παρατηρητές μας εκεί και νομίζω ότι αυτή η παρουσία ήταν θετική για όλο το σώμα. Σούλτς Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να πω στην επικεφαλή της αντιπροσωπής παρατήρησης ότι την ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενημερωτική έκθεση που μας έκανε για την παρατήρηση εκλογών στη Μολδαβία. Γιατί χάρη σε αυτήν την ενημέρωση μάθαμε ότι οι μολδαβικές εκλογές έγιναν με ομαλό και τακτικό τρόπο και με συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ποιο ήταν το πολιτικό κλίμα στη χώρα αυτή. Οι διαδοχικές προεκλογικές εκστρατείες οδήγησαν σε πόλωση και σε ακαμψία των πολιτικών θέσεων. Υπήρχε δυνατότητα συνεννόησης μεταξύ των αντίπαλων πολιτικών δυνάμεων ώστε να επιδιώξει μια διέξοδος από την αποτελμάτωση. Υπάρχει προθυμία από τις πολιτικές δυνάμεις ε, να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την ε, κινησία και την αδράνεια που έχει χαρακτηρίσει τη χώρα τους τελευταίους μήνες. Διαπιστώσετε κάτι τέτοιο. Κυρία Μακοβέ, έχετε το λόγο για τα συμπεράσματα. During the campaign, the, the... Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ε, ακούστηκαν ε, διάφορες ε, επιθετικές παρατηρήσεις, επιθετικές εντός εισαγωγικών. Είναι λογικό σε μια προεκλογική εκστρατεία, υπάρχουν τέτοιες αντιπαραθέσεις πολιτικές, αλλά είναι κάτι το φυσιολογικό σε μια προεκλογική εκστρατεία και η θέση, η παρουσία των πολιτικών ομάδων στα μέσα μαζική ενημέρωση ήταν πολύ ισορροπημένη όπως δήλωσαν και όλες οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που γενικώ είναι αυστηρέ σε τέτοιου είδου αξιολογήσεις. Φαίνεται ότι είναι δυνατό τα τρία δημοκρατικά κόμματα που θα συστήσουν την κυβέρνηση θα σχηματίσουν τον κυβερνητικό συνασπισμό και αν θέλουν να διορίσουν πρόεδρο και να αποφύγουν προώρες εκλογές, είναι υποχρεωμένα να έχουν κάποιες συνομιλίες και να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις και προς το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και συμφωνώ με τον Γκράχαμ ότι θα πρέπει να δούμε και τα μηνύματα που έστειλαν η Λέιδη Άστον και ο Επίτροπος Φίλε. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που εκπροσωπούνται στη Βουλή, ε, καλό θα ήταν ε, να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να βρουν έναν τρόπο ε, για να μην υπάρξει σύγκρουση στο θέμα των προεδρικών εκλογών. Υπάρχει μια σαφής υποστήριξη προς τις δημοκρατικές δυνάμεις. Απ' την άλλη θα πρέπει να συνεργαστούν τα κόμματα για να βρουν μια λύση. Είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε λοιπόν τις εξελίξεις και να δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενο αυτής της συνεννόησης, της συμφωνίας, ποια θα είναι τα όρια αυτής της συμφωνίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλώς, δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, οπότε λύεται η συνεδρίαση.